Dear colleagues, can you please take Αγαπητοί συνάδελφοι, μήπως μπορείτε να καθίσετε γιατί θέλουμε να αρχίσουμε. Μήπως. Uh, so can we... Λοιπόν, μπορεί κανείς να κλείσει την πόρτα παρακαλώ για να αρχίσουμε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Θα αρχίσω με την πληροφόρηση. Ε, υπάρχει αναμετάδοση στο δίκτυο της συνεδρίασης και υπάρχουν και ορισμένες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη. Δηλαδή, ο Υπουργός κ. Μιχαήλ Χρυσοχοίδης που είναι υπεύθυνος για την ανταγωνιστικότητα και την αυσιπλοεία στην Ελλάδα θα ε, μπορούσε να έρθει μόνο σήμερα και όχι αύριο, γι' αυτό αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη και μεταφέραμε το σημείο του το αυριανό κανονικά ως δεύτερο σημερινό. Θα συνεδριάσουμε όσο χρειαστεί, αλλά νομίζω ότι μία ώρα, μία ώρα και ένα τέταρτο για τη συνάντηση αυτή θα αρκούσε. Επίσης θέλω να σας πληροφορήσω ότι η έκθεσή μας για την επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα δυστυχώς αύριο μόνο μπορεί να συζητηθεί γιατί η πρόεδρος της ομάδας που πήγε στην, στην Ελλάδα, ο Βανίς δεν θα είναι σήμερα εδώ. Άρα δεν θα μπορέσει να συζητήσει με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση για τις αλλαγές αυτές, Μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεύτερον, δεύτερο σημείο. Ανακοινώσεις της Προεδρού. Μία ανακοίνωση υπάρχει. Θα την κάνω όταν συζητήσουμε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο. Και επομένως περνάμε τώρα στο 2α που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Τον καλωσορίζω ολόψυχα και θα ήθελα τον συγχαρώ που διατήρησε τη θέση του σε αυτή τη νέα κυβέρνηση στην οποία δόθηκε από ό,τι μαθαίνω ψήφος εμπιστοσύνης με μεγάλη πλειοψηφία του ευχόμαστε καλή επιτυχία και θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι όπως φαντάζεστε γενικότερα στο Κοινοβούλιο εμείς τονίζουμε κυρίως τα μακροοικονομικά στοιχεία, τα προβλήματα γενικότερα της Ευρωζώνης, την κρίση των κρατικών χρεών και δεν ασχολούμαστε στην Περιφερειακή ε, Επιτροπή στη συζήτηση όσο θα έπρεπε τουλάχιστον για την ανάπτυξη και την αναθέρμανση χωρών όπως η Ελλάδα αλλά πιστεύουμε ότι αν δεν υπάρξει επιστροφή στην ανάπτυξη δεν θα μπορέσει η Ελλάδα να αναθερμάνει την οικονομία της και τα δημοσιονομικά της. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε κι εσείς πώς βλέπετε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν στο μέλλον για την ανάπτυξη και την επιτυχία των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα θα ακούγαμε με μεγάλο ενδιαφέρον ότι έχετε να μας πείτε. Θα υπάρξει και χρόνος για ε, ερωταπαντήσεις. Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ μου. Ευχαριστώ πολύ, Δανούτα. Της Επιτροπής, κυρία Χούμπνερ, κύριε Αντιπρόεδρη, ε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ και εδώ και 20 μήνες η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. Μια κρίση στην οποία μας οδήγησε ο εκτροχιασμός του δημοσίου χρέους και η επιδείνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά τη διετία 2007-2009. Μια επιδείνωση που προκλήθηκε αφενός μεν από την παγκόσμια οικονομική κρίση όσο φυσικά και από τις αστοχίες της ίδιας της οικονομικής πολιτικής στην ελληνική οικονομία, στο νέο μακροοικονομικό περιβάλλον που δημιούργησε η Ευρωζώνη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όποιες αστοχίες πολιτικού, πολιτικής δεν αφορούν στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Και θέλω να ευθύς εξ αρχής να επισημάνω ότι στο ευρώ η Ελλάδα μπήκε με μεγάλες προσπάθειες και μεγάλες θυσίες που έκανε ο ελληνικός λαός στη δεκαετία του 90. Οι σκιές που κατά καιρού αφήνονται από μερίδα του πολιτικού κόσμου στην Ευρώπη είναι αβάσιμες, είναι διαλυτικές για την ε, συνοχή της Ευρωζώνης και είναι κατά των ευρωπαϊκών θεσμών και επαναλαμβάνω και πάλι ότι η προσπάθεια που έγινε εκείνη την εποχή της δεκαετίας του 90 ήταν πρωτοφανής. Εγώ προσωπικά ήμουν υφυπουργό σε θέματα αγοράς. Παρέλαβα όταν ορίστηκα υφυπουργό τον πληθωρισμό στο 15% και όταν μπήκαμε στο ευρώ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν μόλις 2%. Σήμερα Βέβαια το διακύβευμα είναι διαφορετικό. Να σώσουμε τη χώρα και να τη βάλουμε ξανά σε τροχιά ανάκαμψης, ισχυροποιώντας τη θέση της Ελλάδος εκεί που δικαιωματικά της ανήκει, στο σκυρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Ξεκινήσαμε πριν από 1,5 χρόνο μια μεγάλη προσπάθεια με το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Μια προσπάθεια ένα πρόγραμμα με δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, τη δημοσιονομική εξυγίανση με μείωση των ελλημάτων και αύξηση των εσόδων και δεύτερον, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών. Μέχρι στιγμής στην Ελλάδα και στα δύο αυτά μέτωπα έχει συντελεστεί σημαντική δουλειά και σπουδαίο αποτέλεσμα. Μια πρόοδος η οποία όμως απέτησε και εξακολουθεί να απαιτεί θυσίες από τον ελληνικό λαό. Τους εργαζόμενους στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία. Μια πρόοδος η οποία ωστόσο έχει προκαλέσει σημαντικά ρήγματα στην κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα και έλλειμμα εμπιστοσύνης στην πολιτική και τους θεσμούς. Και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα είναι σπουδαία γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που να μείωσε το έλλειμμα πέντε ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 12 μήνες. Υπάρχει άλλο κράτος μέλος στην Ευρωζώνη που μείωσε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 50% και να διατηρεί συνθήκες ομαλής λειτουργίας και οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Μεταρρυθμίσαμε το συνταξιδοτικό σύστημα, κάναμε την αγορά εργασίας πιο ευέλικτη, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς μεγάλες, πολύ μεγάλους κοινωνικούς τριγμούς. Λοιπόν, εδώ έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά και αυτό ζητάμε από εσά την αναγνώριση και τίποτα, παραπέ... τίποτε άλλο, τίποτα επιπλέον. Όχι γιατί είναι μια ηθική επιταγή, αλλά γιατί έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα και επαναλαμβάνω με θυσίες του ελληνικού λαού. Αγαπητοί συνάδελφοι στο Ευρωκοινοβούλιο, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα υπάρχει εδώ και δύο εβδομάδες, όπως είπε η κυρία Χούπνερ προηγουμένω, μια νέα κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, μια νέα κυβέρνηση συνεργασίας με σαφή στόχευση. Να εξειδικεύσει και να εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Συνεχίζεται ταυτόχρονα η μεταρρυθμιστική πολιτική που ξεκίνησε εδώ και 1,5 χρόνο με στόχο την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας. Θέλω σήμερα ενώπιόν σας να σταθώ και να σας ενημερώσω διεξοδικά για αυτή την πολιτική που προτάσει πάνω απ' όλα την αναστήλωση της πραγματικής οικονομίας τη μετάβαση από μια εικονική πραγματικότητα σε μια οικονομία παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική. Η Εθνική Στρατηγική Αναπτυξιακής Αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας συνοψίζεται στις ακόλουθες προτεραιότητες και τα εξής πολύ πρακτικά βήματα. Πρώτη προτεραιότητα είναι η εξωστρέφεια η βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, να γίνει η Ελλάδα μια εξωστρεφής οικονομία. Δεύτερο βήμα είναι η επανεξέταση όλων των επενδυτικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια και την οικονομική αποτελεσματικότητα. Ψηφίσαμε πέρυσι και ήδη εφαρμόζουμε έναν νέο σύγχρονο επενδυτικό νόμο με έμφαση στις φοροαπαλλαγές και λιγότερο στις επιδοτήσεις, στροφή προς την τεχνολογία, την εξωστρέφεια, την παραγωγή, την καινοτομία και την νεανική επιχειρηματικότητα. Το τρίτο βήμα ήταν η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού με εθελοντικές μειώσεις τιμών από την πλευρά των επιχειρήσεων στα είδη βασικής διατροφής και κατανάλωσης και τις στοχευμένες παρεμβάσεις κάθε φορά που διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά. Το τέταρτο βήμα ήταν η επιτάχυση της απορρόφησης των πόρων των κοινοτικών προγραμμάτων συνοχής του ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων συνθήκων που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Το πέμπτο βήμα ήταν η αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνη και η εμπέδωση συνθήκων διαφάνειας ώστε να επανακάμψει το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την ελληνική οικονομία. Ένα τέτοιο μέτρο ήταν το fast track που ήδη εξετάζει μια σειρά από μεγάλες επενδύσεις και άλλες πρωτοβουλίες. Το έκτο βήμα ήταν η ψήφιση και εφαρμογή ριζικών διαρθρωτικών αλλαγών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Χτες, χτες μόλις ανακοινώσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραμμα Ελλάδα φιλική προς τις επιχειρήσεις που στόχο έχει την ριζική απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος από τη γραφειοκρατία. Το έβδομο βήμα ήταν η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αποκατάσταση συνθήκων υγιούς ανταγωνισμού σε μια σειρά από αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Το 8 βήμα υλοποιείται αυτή την περίοδο και αφορά στην αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την εξασφάλιση μακροχρόνιας αναπτυξιακής χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Η στρατηγική αυτή, τα οχτώ δηλαδή βήματα αυτά, έχουν αποδώσει τα εξής μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Πρώτον, υπάρχει σημαντική και συνεχιζόμενη αύξηση των μεταποιητικών προϊόντων. Θέλω να σας πω ότι η αύξηση των εξαγωγών χρόνο με το χρόνο στην Ελλάδα είναι της τάξης του 40 περίπου της 100 τον μήνα Οκτώβριο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Και τα ελληνικά προϊόντα απευθύνονται σε αγορές εξαιρετικά απαιτητικέ, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, σε αγορές κυρίως της κεντρικής Ευρώπης και χώρες της Ευρωζώνης. Δεύτερον, υπάρχει αποκλιμάκωση του δίκτυ τιμών καταναλωτή παρά τις ασταθείς συνθήκες στις διεθνείς αγορές των πρώτων υλών και την αύξηση του πληθωρισμού στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Τρίτον, έχει επιτευχθεί μια ριζική αναθεώρηση και αύξηση των ρυθμών απορρόφησης των κοινωτικών πόρων μετά και τη μείωση της εθνικής συμμετοχής. Τέταρτον, Υπάρχει βελτίωση των θεσμικών συνθήκων για την επιχειρηματικότητα και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων με την ίδρυση των υπηρεσιών One Stop Shop. Πέμπτον, έχει ενισχυθεί το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την ελληνική οικονομία και διακρατικές οικονομικές σχέσεις που υποστηρίζουν με γραμμές χρηματοδότησης τις επιχειρήσεις και άλλες διευκολύνσεις σε αυτή την προσπάθεια. Έκτον, έχει δρομολογηθεί η τροποποίηση των κοινοτικών κανονισμών, όπως ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, με πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου, που θα επιτρέψει τη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αναπτυξιακών έργων υποδομής. Έβδομον, 12 μήνες μετά την εξαγγελία για την κατάρτιση του νέου επενδυτικού νόμου ολοκληρώνονται με επιτυχία δύο προκηρύξεις επενδυτικών σχεδίων με διαφάνεια, ενημέρωση του Κοινοβουλίου και απόλυτη τήρηση των προθεσμιών και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο προκηρύξεις. Σε συνθήκες επαπειλούμενης χρεοκοπίας, ο νέος επενδυτικός νόμος έχει υποδεχθεί αθρηστικά στις δύο προκηρύξεις επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Επίσης, στις στοχευμένες επενδυτικές ενισχύσεις καταγράφεται ικανοποιητική συμμετοχή με αποτέλεσμα αυτές οι προκηρύξεις να λειτουργούν ανταγωνιστικά και να βελτιώνεται η ποιότητα των επενδυτικών σχεδίων. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη στρατηγική τόνωση των επενδύσεων και της ανάπτυξης κομβικό ρόλο έχει η προσπάθεια για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα. Μια προσπάθεια με διπλό στόχο. Αφενός με να απλοποιήσει και να αποκεντρώσει τη διαχείριση, να μειώσει τις περιττές διοικητικές διαδικασίες και να ανασυντάξει το στελεχειακό δυναμικό, έτσι ώστε να αυξήσουμε τους ρυθμούς απορρόφησης αφετέρου να απεγκλωβίσουμε πόρους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ που λίμναζαν σε νεκρά έργα και σε νεκρές εκχωρήσεις και να τους προωθήσει σε νέα χρήσιμα έργα για την περιφερειακή οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Σήμερα λοιπόν, Νοέμβριος του 2011, οι εντάξεις έργων είναι στο 92%. Οι νομικές δεσμεύσεις, δηλαδή οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, είναι της τάξης του 53,2%. Και η απορρόφηση είναι στο 26%. Μετά από 21 μήνες καταφέραμε να πάμε τις εντάξεις έργων, τις συμβάσεις και την απορρόφηση 9 φορές παραπάνω. Η δυναμική του προγράμματος φαίνεται και από τα παρακάτω στοιχεία. Θα σας πω για το τελευταίο εξάμεινο οι εντάξεις νέων έργων το τελευταίο εξάμεινο ανέρχονται σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ενεργές συμβάσεις ανέρχονται πλέον σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ από μηδενικές που ήταν πριν από δύο χρόνια περίπου η απορρόφηση του τελευταίου τετραμήνου Ιούνιος-Οκτώβριος του 2011 συγκριτικά με την περσινή του 10 το τετράμινο του 10 Ιούνιος-Οκτώβριος όπως προκύπτει από τα επίσημα αιτήματα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυξημένα κατά 38,3%. Η βελτίωση της διαχείρισης του προγράμματος είναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης που καταγράφει, αξιολογεί ένα προς ένα τα έργα. Υπάρχουν τα 100 έργα σημαίες στο οποίο έχει αναφερθεί επανειλημμένα ο πρόεδρος της Επιτροπής Μπαρόζο και τα έργα ορόσημα σε όλη τη χώρα που θα δώσουν πνοή ξανά στην περιφέρεια. Στόχος είναι να προωθηθούν χρήσιμα έργα υποδομές για τους πολίτες που θα κινήσουν ξανά την αναπτυξιακή διαδικασία αλλά θα δώσουν και λύσεις και ανακούφιση στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα και είναι ακόμα μεγαλύτερο γιατί δυστυχώς επικεντρώνεται η ανεργία στους νέους όπου το ποσοστό αγγίζει τα όρια της ντροπή του 45%. Στην προσπάθεια αυτή που περιέγραψα προηγουμένως συμμετέχει και παρακολουθεί ο Επίτροπος ε, κύριος Χάν και η Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής την οποία θέλω τα στελέχη της οποίας, τον Επίτροπο και τα στελέχη της οποίας θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμβολή τους την πολύτιμη συνεργασία τους και τη βοήθειά τους τα στελέχη της Task Force, τον κύριο Ράιχεμπαχ και τους συνεργάτες του και φυσικά ο ίδιος ο πρόεδρος Μπαρόζο. Για να συνεχιστεί η σημερινή δυναμική υλοποίηση του προγράμματος, εφαρμόζουμε πλέον ένα σύστημα παρακολούθησης, επίτευξης στόχων απορρόφησης, αναεπιχειρησιακό πρόγραμμα και αναέργο. Τέλος, επιτρέψτε μου να σταθώ σε ένα καυτό ζήτημα, ιδιαίτερα μεγάλο ζήτημα που έχει σχέση με την πραγματική μας οικονομία και ειδικότερα σχετίζεται με τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το θέμα της ρευστότητας. Αντιμετωπίζουμε ένα ασφικτικό πρόβλημα ρευστότητας για τη χρηματοδότηση των δανειακών αναγκών των επιχειρήσεων. Και θέλω να σας πω ότι καθημερινά εγώ ως υπουργό αρμόδιος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, βλέπω μπροστά στα μάτια μου να πεθαίνουν και να βγαίνουν από την αγορά επιχειρήσεις υγιέστατες. Γιατί πολλές φορές δεν μπορούν να, πάνουν, να πάρουν ούτε ένα αλέτερο φιντέντ, μια εγγυητική επιστολή. Γιατί πολλές φορές δεν έχουν τη δυνατότητα οι εξαγωγικές μας επιχειρήσεις να πάρουν λίγα χρήματα, μια μικρή προκαταβολή προκειμένου να αγοράσουν τις πρώτες τους ύλε. Και εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και αυτή τη στιγμή μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως την ε, DG Regio κινούμαστε προς τις εξής κατευθύνσεις. Πρώτον, βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση του κανονισμού εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων και στις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ για κεφάλαια κίνησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Να δώσουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν στοιχειοδός ένα κεφάλαιο κίνησης για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους. Δεύτερον, δημιουργούμε ένα εγκυρωτικό ταμείο 500 εκατομμυρίων και πλέον ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τις ελληνικές τράπεζες με αποκλειστικό προορισμό τη χρηματοδότηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης πάντα σε συνεργασία με την Επιτροπή αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή επιχειρούμε είναι ότι προτείνεται η αλλαγή του σχετικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα εγγυητικό ταμείο περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ με πόρους από το ΕΣΠΑ, από το Κοινοτικό Πρόγραμμα Συνοχής της Ελλάδας προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τα μεγάλα έργα, τους δρόμους, τη διαχείριση των σκουπιδιών και άλλες δραστηριότητες τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα και για την ανάπτυξή της και για να λύσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα και για να δημιουργήσει μεγάλα έργα υποδομής αλλά και για να καταπολεμήσουμε το οξύ πρόβλημα της ανεργίας που περιέγραψα προηγουμένως. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κλείνοντα θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τη συμμετοχή σας σε αυτήν την συνάντησή μας εδώ, την οποία διοργάνωσε η κυρία Χούπνερ. Να σας διαβεβαιώσω ότι και πάλι ότι στην Ελλάδα γίνεται μια πολύ μεγάλη υπεράνθρωπη σκληρή προσπάθεια με θυσίες του ελληνικού λαού για να κάνουμε τη χώρα μας και την ελληνική οικονομία παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική. Εργαζόμαστε σκληρά για να αναστηλώσουμε την πραγματική οικονομία, δίνοντας έμφαση στην πραγματική οικονομία, στην εργασία και στην ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάδα βάζει τις βάσεις, μέσα στην κρίση αυτήν, βάζει τις βάσεις ενός νέου προτύπου, ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Χρειάζεται να γίνουν θυσίες περαιτέρω, να υλοποιηθούν σκληρές αποφάσεις, να αλλάξουν νοοτροπίες ετών, με επίπονες προσπάθειες διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις, ώστε να φέρουμε την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Ταυτόχρονα Χρειαζόμαστε όλοι στην Ευρώπη να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, μιας και η κρίση αποκτά ευρύτερα χαρακτηριστικά. Η επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης είναι μια πρόκληση για όλους μας. Η επιτυχής αντιμετώπιση αυτή της, πρόκλησης πρέπει να γίνει με όρους συνεργασίας και αλληλεγγύης όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, thank Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Θερμά ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνετε και φαντάζομαι ότι η πρόκλησή σας είναι όχι μόνο να επανέλθει στο δρόμο της ανάπτυξης η Ελλάδα, αλλά να αλλάξουν θεμελίων πολλά πράγματα και να βάλετε τις βάσεις για μια υφόρο ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μπορούμε τώρα να προβλέψουμε ένα χρόνο για συζήτηση και αφού με τους συναδέλφους θα δώσω το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για σύντομα σχόλια. Πρώτη η Κωνσταντζα Κρέλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, η Περιφερειακή Επιτροπή ε, ανέκαθεν ε, προσπαθούσε να κάνει το καλύτερο για την Ελλάδα. Αυτά που είναι εφικτά να τα στηρίξει έτσι ώστε να επιτευχθεί η διαρθρωτική αλλαγή και έτσι ώστε πραγματικά να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η δική σας η χώρα πράγματι καταβάλει αυτή τη στιγμή τεράστιες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες και γνωρίζουμε επίσης ότι οι Έλληνες πολίτες ε, καταβάλουν τεράστιες θυσίες. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά και επιτρέψτε μου να επανέλθω σε ένα θέμα που θίξατε εσείς. Δηλαδή, αυτές ε, η χρήση των διαρθρωτικών κονδυλίων με ποια ταχύτητα, πόσο γρήγορα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι απτά και ορατά. Και επίσης, αυτή η κατάσταση, αν υποθέσουμε ότι βελτιώνεται, θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην αγορά εργασίας και πόσο γρήγορα. Μήπως έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα για επενδύσεις που γίνονται ή θα μπορούν να γίνουν στο μέλλον. Ξέρετε, τα λέω όλα αυτά γιατί εγώ ε, συμμετείχα σε αυτή την αντιπροσωπεία η οποία επισκέφτηκε τον Ιούλιο την Ελλάδα και στην Ελλάδα επιτόπου ενημερωθήκαμε για το ότι η κυβέρνηση κατέβαλε μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αποκέντρωσης κυρίως για τη χρήση των διαρθρωτικών κονδυλίων. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Όμως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υλοποιούνται τα προγράμματα που είχαν προβλεφθεί στο πλαίσιο της διαρθρωτικής πολιτικής. Και ρωτώ τώρα, Ποια ακριβώ είναι η κατάσταση. Είσαστε αναγκασμένοι να ανακαλέσετε όλα τα προγράμματα ή μήπω συνεργάζεστε επί τη ουσία με τι περιφέρειες. μπορείτε λιγάκι να μα εξηγήσετε αυτό το θέμα τη περιφερειακή συνεργασία και χρήση κονδυλίων. Να ακούσουμε και μερικέ άλλε ερωτήσει. Ο Ευγένη Κυρίλοφ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε και σας, κύριε Υπουργέ. Ε, χαιρόμαστε για την παρουσία σας εδώ είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και η συζήτηση των προβλημάτων. Και αυτό όχι μόνο για χάρη της Ελλάδας. Γιατί τι σημαίνει συνοχή. Συνοχή σημαίνει αλληλεγγύη σε τελική ανάλυση. Και στην Επιτροπή μας είμαστε ανέκαθεν υπέρ τέτοιων πολιτικών ενεργών, ιδιαίτερα προς χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι ότι δεν πρόκειται να ξεφορτωθούμε γρήγορα την κρίση. Όπως λέει και μια αμερικανική ε, φράση, μην ανησυχείτε, για μια δεκαετία θα την έχετε ακόμη. Και ακούσαμε για αυτή τη φοβερή έλλειψη ρευστότητα, για την ε, απώλεια των μικρομεσών επιχειρήσεων και ότι ούτε κάνει η αύξηση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής δεν βοηθάει στην ανάπτυξη. Και αυτό μας δίνει κάποια επιχειρήματα για τους μελλοντικού προπολογισμού. Γιατί η λιτότητα δυστυχώ σκοτώνει τους πάντες, όχι μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν δεν ε, εφαρμοστεί με το σωστό τρόπο. Γιατί παρά τη λιτότητα το έλλειμμα σας αυξάνεται παρά τα σωστά μέτρα, τα δρακόντια μέτρα λιτότητας και προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα λοιπόν από αυτήν την άποψη να σας θέσω μια ερώτηση γιατί πολύ πιθανό πολλές χώρες να χρειαστεί να διδαχθούν διάφορα πράγματα από την ε, στιγμή αυτή κρίση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Στρατηγικής και τον προγραμματισμό, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε και πώς μπορείτε να βοηθήσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί μαζικά εξαφανίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες. Ε, χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη για να προχωρήσουν οι μικρομεσαίες και δυστυχώς τέτοια ανάπτυξη δεν υπάρχει πουθενά. Σας ευχαριστούμε πάντως που ήρθατε. Επαναλαμβάνω, τα προβλήματα αυτά δεν είναι μόνο χαρακτηριστικά προβλήματα της Ελλάδος, είναι δυστυχώς προβλήματα ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ακούσουμε ακόμη έναν ομιλητή, τον κύριο Τρεμόπουλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, προφανώς βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση του συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η Ελλάδα έχει τις δικές της αδυναμίες, για να το πούμε κομψά, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με μια λάθος συνταγή τα το, το τελευταία δύο χρόνια. Με δεδομένο ότι την ύφεση που για πέντε συνεχόμενα χρόνια έχει η Ελλάδα εξαιτίας της ακολουθούμενης πολιτικής, εξαιτίας της πολύ μεγάλης μείωσης του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και την πολύ χαμηλή απορροφητικότητα 23% του ΕΣΠΑ μέχρι τώρα, θα ήθελα συγκεκριμένα να μας πείτε τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα, ούτως ώστε να μπορεί να ελπίζει κανείς ότι θα υπάρξουν άλλα αποτελέσματα. Δεύτερο, με ποιες προτάσεις συμμετείχε η Ελλάδα στη συζήτηση για τη νέα πολιτική συνοχή μετά το 2014. Έχει εξασφαλιστεί μετά από δημόσια διαβούλευση μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική υποστήριξη. Και τρίτον, με ποιο τρόπο υποστηρίζεται τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου προγραμματικού πλαισίου. Μένω σε αυτά που είναι το αντικείμενο της Επιτροπής αυτής. Maybe you comment on πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε στους τρεις ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ. Τα προγράμματα τα διαρθρωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλω να σας πω ότι ε, δεν είναι προγράμματα τα οποία τρέχουν γρήγορα. Βλέπετε σε όλες τις χώρες υπάρχουν προβλήματα απορρόφησης. Θα έλεγα ότι είναι μεσοπρόθεσμης απόδοσης προγράμματα με πολλές διαδικασίες και στην Ελλάδα ε, έχουμε ακόμα περισσότερα προβλήματα λόγω των, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή με τον κρατικό μηχανισμό και τη δημόσια διοίκηση. Ωστόσο, αυτό το οποίο κάναμε τον τελευταίο καιρό, με την βοήθεια και τη συνεργασία της Επιτροπής και την αλλαγή μιας σειράς κανόνων οι οποίοι υπήρχαν στην αξιοποίηση, στη χρήση και τη διαχείριση των κοινωνικών πόρων και τώρα αλλάζουν ριζικά, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, αν θέλετε. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα, είχαμε περιπτώσεις καταρχήν είχαμε περίπου 5 δισεκατομμύρια έργα νεκρά, δηλαδή τα οποία δεν είχαν ξεκινήσει ποτέ. Αυτά τώρα πια έχουν μείνει ελάχιστα. Σας είπα ότι το πρόγραμμα έχει πλέον, είναι ενταγμένα ζωντανά έργα 92%. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχαν φαινόμενα πολλών εκχωρήσεων. Δηλαδή το Υπουργείο στην Περιφέρεια, η Περιφέρεια στο Δήμο, ο Δήμος σε κάποιο άλλο, σε ένα πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά έχουν καταργηθεί, έχουν τελειώσει. Και έτσι επιτρέπεται μόνο μία εκχώρηση και αυτό καθιστά την απορρόφηση και την ορίμανση των ε, projects πιο γρήγορη. Έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες με αποτέλεσμα να είμαστε εμείς ήδη πιο αποτελεσματικοί στην απορρόφηση. Επίσης, θέλω να σας πω ότι πάλι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Regio, έχουμε δημιουργήσει ένα στρατό από υπτάμενους τεχνικούς, συμβούλους οι οποίοι τρέχουν σε όλη τη χώρα, ακόμα και στους πιο μικρούς δήμους της χώρας, προκειμένου να οριμάσουν γρήγορα τα έργα. Σας λέω πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και αποδίδουν προς την κατεύθυνση του αποτελέσματος που σας ανέφερα προηγουμένως. Άρα λοιπόν είναι εξασφαλισμένο πλέον ότι από εδώ και πέρα ε, όλη αυτή η διαδικασία της απορρόφησης του προγράμματος θα τρέξει, άρχισε ήδη τρέχει και θα τρέξει με μεγαλύτερους ρυθμούς. Εάν ε, με ρωτήσετε εάν ε, συμβάλλει η απορρόφηση των κοινοτικών πόρων στην αγορά εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα. Να σας πω ένα παράδειγμα λοιπόν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αναστολή πέντε μεγάλα οδικά έργα, κατασκευή δρόμων δηλαδή, τα οποία δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του δημοσίου και των εργολάβων μεταξύ των δημοσίων, των εργολάβων και των τραπεζών που συμμετέχουν. Είναι έργα παραχώρησης. Είναι έργα αξίας περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εάν με την προσπάθεια που κάνουμε στην Επιτροπή τώρα και στην Task Force ξαναρχίσουν αυτά τα έργα σε λίγους μήνες, θα έχουμε περίπου 10.000 θέσεις εργασίας που θα ξεκινήσουν αμέσως να λειτουργούν. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μια χώρα η οποία ξεπερνάει τώρα πια το 20% στην ενεργεία. Σε ό,τι αφορά το, το δεύτερο ερώτημά σας, νομίζω ότι μέρα με τη μέρα πράγματι το πρόβλημα εξαπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Ακόμα και χώρες που δεν, έχουν, που δεν αντιμετωπίζουν δημοσιονομικό πρόβλημα υπάρχει το πρόβλημα, ένα πραγματικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Και είναι το πρόβλημα της ύφεση. Και η ύφεση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των λαών και των εθνών και των χωρών μας. Γιατί είναι η αιτία που δημιουργεί ανεργία, είναι η αιτία που δημιουργεί έλλειψη πλούτου, είναι η αιτία που δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα. Άρα λοιπόν την ύφεση αυτών των εχθρών πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Παλεύοντας ταυτόχρονα τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλά μόνο με τη δημοσιονομική σταθερότητα, χωρίς αναπτυξιακές πολιτικές, δεν τα πουθενά. Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα της χρήσης των κοινωτικών πόρων το πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε πώς θα τους καταστήσουμε περαιτέρω δύο πράγματα. Το ένα πιο αποτελεσματικούς για να τονώσουν την οικονομία αλλά και κάτι άλλο πιο χρήσιμους και εννοώ πιο χρήσιμους κατά τη γνώμη να δούμε το θέμα της λεγόμενης επιλεξιμότητας eligibility να δούμε το θέμα της επιλεξιμότητας διότι η επιλεξιμότητα εφόσον επικεντρωθεί, είναι στοχευμένη σε συγκεκριμένες δράσεις της οικονομίας, ανάλογα με τα συγκριτικά πλονεκτήματα που διαθέτει κάθε χώρα και η κάθε οικονομία, τότε λοιπόν οι πόροι θα γίνουν ακόμα αποτελεσματικότεροι και ακόμα χρησιμότεροι. Στην Ελλάδα προσπαθούμε να, επειδή με ρωτάτε, Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με πάρα πολλούς τρόπους έτσι ώστε τουλάχιστον αυτές οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης εξωστρεφούς και βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης να τη στηρίξουμε. Θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα. Έχουμε 2.000 εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν εξαγωγές ύψους 20 περίπου τώρα δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή το 10% του ΑΕΠ της χώρας. Πριν από λίγες εβδομάδες εκπονήσαμε ένα πρόγραμμα και στηρίζουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις εξαγωγικές με ένα ειδικό πρόγραμμα μαζί με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων ούτω ώστε να μην υπάρξει καμιά επιχείρηση εξαγωγική στη χώρα που δεν θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει πρώτες ύλε ή τα υλικά που χρειάζονται προκειμένου να εκτελέσει τις παραγγελίες της προς τους πελάτες του εξωτερικό. Αυτό είναι μια σημαντική συμβολή. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα παραδείγματα γιατί προσπαθούμε να υποκαταστήσουμε το τραπεζικό σύστημα το οποίο δυστυχώς αυτή τη στιγμή για τους γνωστούς συστημικούς λόγους δεν λειτουργεί. Τέλος, πράγματι στην Ελλάδα έχουμε μια σημαντική μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων λόγω του προγράμματος σταθεροποίησης και προσαρμογής που εφαρμόζουμε. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στην, στα ήδη μειωμένα κονδύλια που διαθέτουμε και στην ανάπτυξη της χώρας το υπερβαίνουμε πια αυτό το πρόβλημα σε λίγο επειδή η σχέση κοινοτική συμμετοχής και εθνικής συμμετοχής ουσιαστικά με το 95-5 μηδενίζεται η εθνική συμμετοχή. Άρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε την εθνική προσπάθεια που κάνουμε για την ανάπτυξη και τις υποδομές μέσα από αυτήν τη νέα σχέση η οποία διαμορφώνεται στο, στα προγράμματα της ε, συνοχής της χώρας μας. Ε, εμείς θα κάνουμε πράγματι ετέθη ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για την πολιτική συνοχή. Είναι κρίσιμο ζήτημα για όλους μας. Θα κουβεντιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και στο Συμβούλιο Συνοχής, των Υπουργών της Συνοχής. Νομίζω ότι πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις που απαντάνε στις ανάγκες της συγκυρίας. Εμείς θα ανοίξουμε ένα διάλογο με τους φορείς, τα κόμματα, και όλους τους αρμόδιους στην Ελλάδα έτσι ώστε ε, οι προτάσεις μας να απαντούν στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό βεβαίως εντάσσεται και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης μιας και φέτος για δεύτερη χρονιά διαθέτουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας ερετές ε, δευτεροβάθμιες και βέβαια πολύ μεγάλο συνοποιημένους δήμους. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε τρεις ακόμη που ζήτησαν το λόγο. Την κυρία Φαβέλα, Τέλερ και Πέτερ Σίμαν. Η κυρία Φαβέλα πρώτη. Πρόεδρος, κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία στη δουλειά σας. Όλοι οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι το ευχόμαστε αυτό. Κύριε Υπουργέ, είχατε δηλώσει το παρελθόν ότι για την περιφερειακή ανάπτυξη χρειάζονται εμβληματικά έργα. Είπατε ότι όλα αυτά τα έργα, τα παραδοσιακά που είχαμε, συντελούσαν στην ανάπτυξη. Τώρα πρέπει να πάμε σε ρηξικέλευτες προτάσεις για να ε, αναζωπηρωθεί η περιφερειακή ανάπτυξη, οι τοπικές κοινωνίες κτλ. Ε, ένας τέτοιος τομέας είναι η κρουαζιέρα είστε υπεύθυνο και για αυτό το τομέα, όχι μόνο για την περιφερειακή ανάπτυξη. Έξι περιφέρειες της Ελλάδος μπορούν να έχουν home port κρουαζιέρα. Δηλαδή το κρουαζερόπλιο το οποίο έχει από 2.000 μέχρι 6.000 επισκέπτες επάνω μπορεί να ξεκινάει από έξι λιμάνια που καλύπτουν έξι περιφέρειες της χώρας. Αυτό όλοι αντιλαμβανόμαστε τι ευεργετική οικονομική επιρροή έχει και στην περιφέρεια και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό όμως δεν έχει προχωρήσει κύριε Υπουργέ. Υπάρχει το θέμα του καμποτάζ. Για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει. Είναι μια μεταρρύθμιση αυτή την οποία σας υποδεικνύω και δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος. Άρα λοιπόν ούτε γραφειοκρατική διαδικασία μεγάλη χρειάζεται, ούτε οικονομικό κόστος. Είναι μία όμως πάρα πολύ ουσιαστική μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Καταρχήν ε, θα ήθελα να σας καλωσορίσω που ήρθατε εδώ και που θελήσατε να μας παρουσιάσετε τη δουλειά σας και μάλιστα με ειλικρίνεια, με παρησία. Ε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν αποκρύψατε και τις ε, δυσκολίες που αντιμετωπίζετε γιατί είμαι σίγουρος ότι και εσείς είσαστε αναγκασμένος τα λάθη του παρελθόντος να τα διορθώσετε σε ταχύτατο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το στοιχείο, το στοιχείο χρόνος και αυτό αυτό είναι το στοιχείο που με ανάγκασε, με ότισε μάλλον να σας κάνω εξή ερώτηση. Ε, το 2012 τελειώνει η περίοδος, η χρήση και ήδη μιλάμε για την περίοδο 2014 μέχρι το 2020. Έχουν ήδη κατατεθεί κάποια σχέδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούμε φωνές ε, οι οποίες ε, αμφισβητούν την αξία της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής και λένε ότι αν θέλουμε να έχουμε μια περιφερειακή πολιτική αυτή θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερο στοχευμένη και όχι να διασπείρεται σε κράτη και περιφέρειες. Εδώ στην αίθουσα σίγουρα έχετε συμμάχους. Ε, ξέρετε γιατί, γιατί και εμεί θέλουμε να συνεχίσει η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχή να εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση την αρχή τη επικουρικότητα, αλλά και τη αλληλεγγύη. Κατόπιν τούτου φτάνω στην παράκλησή μου. Καταρχήν, αναφερθήκατε σε κάποια μέτρα. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να συνεχίσετε να εφαρμόζετε αυτά τα μέτρα. Από την άλλη βέβαια ακούμε και το είπατε κι εσείς ότι στη χώρα, στην Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στην εφαρμογή αυτών των μέτρων. Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι τόσο μεγάλη η απορροφητικότητα όπως θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό λοιπόν σας ρωτώ, εσείς σκοπεύετε να τα δημοσιοποιήσετε όλα αυτά τα εμπόδια και ε, όχι μόνο να ε, χρησιμοποιείτε τη βοήθεια της Κομισιόν που σας προσφέρετε, αλλά όταν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο, να ζητήσετε βοήθεια και από άλλα κράτη, συγκεκριμένα και μεμονωμένα, έτσι ώστε στο πλαίσιο της αλληλεγγύης τα κράτη αυτά να σας βοηθήσουν για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε την κρίση που μαστίζει τη χώρα σας και να μην ε, καταστεί τελικά, να μην προκύψει ε, αυτή η κατάσταση όπου δεν θα απορροφήσει τα κονδύλια, θα επιστραφούν, θα πάνε πίσω στις ε, χώρες πηγή. Αυτό όμως δεν προωθεί την περιφερειακή πολιτική, ούτε τη διαρθρωτική πολιτική και σε τελική ανάλυση σε συζητήσεις που θα γίνουν στο μέλλον σχετικά με τα μελλοντικά προγράμματα για το 2014 και 2020. Εκεί αν δεν γίνουν όλα αυτά θα αναγκαστούμε να ξανασυζητήσουμε τις προϋποθέσεις. Ο Πέτερ Ζήμων. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα κι εγώ να ε, συνεχίσω με αυτό που τέλειωσε ο κύριος ε, Τσέλερ, δηλαδή τα διοικητικά προβλήματα κατά την χρήση των ε, διαρθρωτικών κονδυλίων, αλλά και στη διοίκηση, στην ελληνική διοίκηση, κάτι που εντοπίστηκε ως πρόβλημα αλλά και ως κλειδί. Το κλειδί που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αν λυθούν αυτά τα διοικητικά προβλήματα. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρελθόν προσφέραμε αρρωγή, βοήθεια, προσφέραμε βοήθεια και στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τους βοηθήσαμε αυτό μέσα από μια εταιρική σχέση, μια σχέση ε, που αφορούσε πόλεις της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, ένα είδος αδελφοποίησης. Πόλεις βοηθούσαν πόλεις στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Και ξέρετε κάτι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που αυτό το πείραμα ε, επισφραγίστηκε, επισ... σφραγίστηκε με επιτυχία, όπου υπάρχουν πολλοί ε, οι οποίες ε, μπόρεσαν σε πάρα πολλούς τομείς ε, να εγκαταστήσουν νέα διοικητικές, νέες διοικητικές δομές και αυτό μέσα από κοινωνικά προγράμματα. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα Τάσης City 10. Σήμερα λοιπόν θέλω να ρωτήσω για τη βελτίωση των διοικητικών δομών. Όταν μιλάμε για βελτίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, Πιστεύετε ότι έχει νόημα να εφαρμοστεί, αν θέλετε, αυτή η ιδέα. Δηλαδή, να υπάρχει στην Ελλάδα, στην περίπτωση της Ελλάδας, συνεργασία μεταξύ πόλεων, πόλη με πόλη. Να είναι, ας πούμε, ένα πρόγραμμα τάσης City Greece. Αδελφοποίηση πόλεων με την Ελλάδα, έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να υπάρξει μία βελτίωση. Ε, Κορνέλια Ένστιν, τελευταία μιλήτρια. Ε, ε, Κοιτάξτε, ε, και εμένα με έτσι, το ότι πολλοί μίλησαν για την ανάπτυξη και για τη διοίκηση. Ίσως λοιπόν πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα προέκυψαν τεράστια κοινωνικά προβλήματα τα οποία επιτάθηκαν λόγω της πολιτικής λιτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου λοιπόν η ερώτηση είναι η εξής κύριε Υπουργέ. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε, κυρίως στον τομέα του ESF, του Εγγυητικού Ταμείου, θα υπάρχουν ε, κάποια χρήματα για την αντιμετώπιση της ε, φτώχειας και άλλων ε, παρεμφερών προβλημάτων. Και η τελευταία μου παρατήρηση είναι η εξή. Το βρίσκω πάρα πολύ καλό που ήρθατε εδώ και μιλήσατε ανοιχτά για τα προβλήματά σας. Γιατί στη τελική ανάλυση η Ελλάδα δεν είναι και η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω κρίσης. κατόπιν τούτου θεωρώ ότι το να μιλάει κανείς ειλικρινά αυτό είναι πάντα σωστό και γι' αυτό κύριε Υπουργέ σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν να πω ότι ξεκινώντας από την ερωτήσει της κυρία Τζαβέλα ε, πρέπει να δούμε από μια νέα οπτική γωνία την αξιοποίηση όλων των πόρων, είτε είναι κοινοτική, είτε είναι εθνική, είτε είναι ιδιωτική, προς την κατεύθυνση της προστιθέμενης αξίας που πρέπει κάθε φορά να έχει μια δράση την οποία κάνουμε. Εάν δεν έχει προστιθέμενη αξία, τότε σημαίνει ότι δεν λειτουργούμε σωστά και ότι οι πολιτικές μας δεν στοχεύουν στην ανάπτυξη, στην πραγματική οικονομία και στην απασχόληση. Άρα λοιπόν ένα κρατούμενο αυτό και αν μιλάμε για τα εμβληματικά έργα, ακριβώς η αποστολή και η ανάδειξη αυτών των εμβληματικών έργων είναι για κάθε περιφέρεια ή για κάθε τομέα αντιστοιχεί ένα εμβληματικό έργο από ένα έως τρία μάλλον εμβληματικά έργα τα οποία σηματοδοτούν ακριβώς αυτή τη στόχευση της προστιθέμενης αξίας στην πραγματική οικονομία, στην εργασία και τελικά το κοινωνικό όφελος. Το... Η κυρία Τζαβέλα έστε στο θέμα της κρουαζιέρας. Πράγματι, τελευταίο καιρό υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει πολλαπλασιασμός των ε, επισκεπτών που επισκέπτονται αυτή τη στιγμή την Ελλάδα με την κρουαζιέρα. Φέτος ήταν μια ιδιαίτερα καλή χρονιά. Η Ελλάδα είναι προσφυλής, δημοφιλής τουρισμός, ε, ε, προορισμός. Ήδη έχουμε προτάσεις για δημιουργία homeport σε, κάποιες, σε κάποια λιμάνια της χώρας, κυρίως στην νησιωτική Ελλάδα και αυτή η υπόθεση πάει εξαιρετικά θετικά. Θέλω λοιπόν να σας ανακοινώσω γιατί συμφωνώ μαζί σας ότι τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε σε κατάθεση διάταξης νόμου προκειμένου να καταργήσουμε πλήρως το καμποτάζ, να απελευθερώσουμε την κρουαζιέρα και αυτό είναι αναγκαίο προκειμένου ο κάθε επιχειρηματίας με βάση και το ισχύον καθεστώς στη χώρα και σε ολόκληρη την Ευρώπη με σεβασμό στο περιβάλλον να προωθεί τις δικές του επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην κατάργηση και την πλήρη άρση του καμποτάζ. Θέσατε οι τρεις τελευταίες ερωτήσεις αφορούσαν τα εμπόδια που υπάρχουν στην επιχειρηματικότητα, τα εμπόδια που υπάρχουν μέσα από τη δημόσια διοίκηση, στην άσκηση και στην εφαρμογή των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Υπάρχουν πράγματι μια σειρά από προβλήματα τα οποία δημιουργούν καθυστερήσεις, αναχώματα, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην υλοποίηση των πολιτικών μας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η Ελλάδα έχει υλοποιήσει τρία κοινωτικά πλαίσια στήριξης, τρία προγράμματα δηλαδή, με πλήρη επιτυχία να είστε βέβαιοι ότι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και θα απορροφηθεί πλήρως. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προβλήματα. Και η περιγραφή των προβλημάτων έχει να κάνει και με τις ανακατατάξεις που πολλές φορές γίνονται όπως έγινε εμάς με το νέο σχέδιο για τις περιφέρειες όπου υπάρχει μια φυσιολογική αναστάτωση με τις εκλεγμένες περιφέρειες όπως επίσης υπάρχουν και τεράστια προβλήματα με τις περικοπές μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Ε, δεν υπάρχει λόγος να κρύβουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Αντιθέτως πρέπει να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να τα λύνουμε από κοινού. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν εργαζόμαστε συστηματικά και τον τελευταίο καιρό έχουμε κάνει μια σειρά από νέους νόμους που απλοποιούμε τις διαδικασίες για το επιχειρήν. Να κάνουμε δηλαδή την Ελλάδα φιλική στις επενδύσεις. Χθες ανακοίνωσα την επέκταση και σε μικρότερες επενδύσεις της διαδικασίας του Fast Track. Δημιουργείται στην Ελλάδα ένα ειδικό κέντρο αδειοδότησης για όλες τις επενδύσεις πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή όποιος θέλει να επενδύσει στη χώρα πάει σε, ένα, σε μια υπηρεσία one-stop shop, καταθέτει το φάκελό του και αυτή η υπηρεσία αναλαμβάνει να διεκπαιρεώσει πλήρως μέχρι αδειοδότησης όλη την επένδυση, όλο το φάκελο. Και όλα αυτά γίνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί θέλω να σας πω και να στείλω ένα μήνυμα εδώ από τη συνάντησή μας εδώ σήμερα, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή επιχειρεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση, μια μεγάλη αλλαγή. Επιχειρούμε να αλλάξουμε ριζικά και την ελληνική κοινωνία και το πολιτικό μας σύστημα, τους θεσμούς, αλλά κυρίως αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε είναι από τη μια μεριά το κράτος και όσες τρευλώσεις αυτό έχει και από την άλλη πλευρά το μοντέλο της οικονομίας για να το καταστήσουμε παραγωγικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό. Για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στην οικονομία, για να δώσουμε δουλειά στους νέους της Ελλάδας. Η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη πρίκα, μια πολύ μεγάλη περιουσία. Και αυτό είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο διαθέτουμε ένα εκατομμύριο περίπου καλά μορφωμένους νέους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αλλά δυστυχώς αυτό το δυναμικό, αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο μαστίζεται αυτή τη στιγμή από ανεργία. Γίνεται λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει ριζικά και το κράτος και το μοντέλο της ανάπτυξης. Και εδώ υπάρχουν συνεργασίες, όπως σας είπα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Task Force, αλλά και πολύ σωστά είπατε, διμερός από άλλες, με άλλες χώρες. Εγώ προσωπικά τον τελευταίο καιρό έχω συνεργαστεί επανειλημμένα με συναδέλφους μου στη Γερμανία, στην Αυστρία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, πάρα πολλές χώρες, προκειμένου να ανταλλάξουμε know-how, εμπειρίες, καλές πρακτικές που θα βοηθήσουν στο να γίνουμε ακόμα περισσότερο αποτελεσματικοί. Και βεβαίως αφορά και την αυτοδιοίκηση αυτό. Βεβαίως η, αδελφοποίηση πόλεων είναι μια διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια άμεση επέμβαση, θα έλεγα, στήριξης και τεχνικής βοήθειας που χρειάζονται οι νέοι μεγάλοι δήμοι και οι περιφέρειες προκειμένου σε πρώτη φάση να απορροφήσουμε το, τους πόρους, να ετοιμάσουμε τα έργα, να τα οριμάσουμε σε μελέτες και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις ανταλλαγές μεταξύ πόλεων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βεβαίως σκεφτόμαστε το νέο ταμείο που αναφέρατε. Είμαι απόλυτα σύμφωνος για το θέμα της φτώχειας ε, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσουμε περαιτέρω το άνεργο δυναμικό της χώρας. Ήδη σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στο χώρο της λεγόμενης κοινωνικής εργασίας, περίπου 50.000 θέσεις. Το λέω ε, γιατί είναι μια υπόθεση που προετοιμάζεται εδώ και αρκετό καιρό θα ξεκινήσει ούτω ώστε να δώσουμε δουλειά έστω για λίγους μήνες, για έξι μήνες σε άνεργους οι οποίοι έχουν απολυθεί από τις επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια προκειμένου να απασχοληθούν και να αποκτήσουν και καινούργιες αν θέλετε εξειδικεύσεις. Κλείνοντας λοιπόν να πω ότι Do we have any other questions? No. Okay. λοιπόν και αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας σε αυτήν την ε, τόσο μαζική συνάντηση και αφού ευχαριστήσω και την κυρία Χούπνερ για την πρωτοβουλία που είχε να οργανώσει αυτή τη συνάντηση, την τόσο χρήσιμη για μας. Ελπίζω να είναι και για σας χρήσιμη μετά τις πληροφορίες που σας ε, μετέφερα εδώ σήμερα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι θυσίε του ελληνικού λαού είμαι βέβαιος ότι με τη δική μας δουλειά θα πιάσουν τόπο. Οι θυσίε του ελληνικού λαού και μετά τη νέα εξέλιξη που είχαμε στον τόπο με την κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης είμαι βέβαιος ότι θα αποδώσουν ακόμα περισσότερο και ότι εν τέλει οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου θα δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα στη χώρα. Δηλαδή μια σταθεροποίηση, και ένα μήνυμα ότι ανοίγει μια νέα περίοδος για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. So if Παρακαλώ και τον ε, κύριο Σαν Μαριζέλερ που είναι υπεύθυνος διευθυντής για τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών και ειδικότερα για την Ελλάδα να μας πει και αυτός δύο λόγια να μας πει τα, τι δουλειά κάνει η Γενική του Διεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, η πολιτική συνοχής είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία σε αυτές τους δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα διαθέτει 2 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή και ένα τέταρτο από αυτά έχουν μόνο απορροφηθεί, 22 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες για να καταπολεμηθεί η ύφεση η Κομισιόν δημιούργησε μία ειδική task force με στόχο να επιταχύνει πράγματι την, αφορόφηση, την απορρόφηση επιτόπου και η task force αυτή θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει για τεχνική υποβοήθηση και χρησιμοποίηση του κοινωνικού ταμείου και των διοικητικών της δυνατοτήτων υποβοήθησης. χρειάζονται βέβαια, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες και την υποστήριξη όλων των κρατών μελών για να υπάρξει μία αμοιβαία πληροφόρηση και βοήθεια. Και τρίτον, να σας δώσω μερικά παραδείγματα της δουλειάς μας. Ο Επίτροπος Χάν προς στιγμήν επικεντρώνεται σε μερικές προτεραιότητες που θα έχουν σχέδια που θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επίπτωση επιτόπου και κάνει ό,τι μπορεί ώστε να εφαρμοστούν με τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία. Για το πρόβλημα της ρευστότητας, τους τελευταίους δύο μήνες, πρώτα πρώτα αυξήσαμε το ρυθμό δανειοδοτήσεων μας στο μέγιστο και γι' αυτό 400 εκατομμύρια παραπάνω δόθηκαν στην Ελλάδα ως πρόσθετη βοήθεια για να λυθεί αυτό το πρόβλημα της ρευστότητας. Επίσης, έχει σχεδόν εγκριθεί και από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να γίνει ένα top-up 10% παραπάνω, ώστε να μπορέσει η Κομισιόν αυτά τα περίπου 400 εκατομμύρια παραπάνω να τα διαθέσει πριν τελειώσει ο χρόνος. Μετά με τη βοήθεια της ΕΤΕ προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να τις βοηθήσουμε στο πρόβλημα ρευστότητάς τους ε, δημιουργώντας ένα ειδικό ταμείο εγγυήσεων και τέλος κάτι όμως που θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο γιατί χρειάζεται αλλαγή του ισχύοντος κανονισμού και σε αυτό θέλουμε και τη δική σας βοήθεια είναι το επόμενο θέμα που προβλέψατε να υπάρξει ένα μεγάλο ταμείο εγγυήσεων που να αντιμετωπίζει ακριβώς τέτοια προβλήματα ρευτότητα. Επίσης προσπαθήσαμε να περισσώσουμε τα κυριότερα μεγάλα συμβόλαια για την Ελλάδα όπως για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε με τις εθνικές αρχές να δούμε πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί ή να ξαναρχίσει ε, το έργο αυτό. Τέλος, θέλω να επιμείνω για το θέμα της διακυβέρνησης, governance. Πρέπει να εξυγχρονιστεί ο δημόσιος τομέας, να είναι πιο αποτελεσματικός, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, και η αρχή της υπευθυνότητας ή της ευθύνης όλων των παραγόντων να είναι πραγματική και να λυθούν και ορισμένες δυσκολίες στο τομέα των δημοσίων προμηθειών, κατάρτισης του κτηματολογίου κλπ. Όλα αυτά υπό τον τίτλο διακυβέρνηση. Κυρία Πρόεδρε, κοντολογής η η πολιτική συνοχή παραμένει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση των τεραστίων δυσκολιών που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Στην Επιτροπή μας όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν να τροποποιήσουμε το συντομότερο δυνατό τον κανονισμό ώστε να επιτρέψουμε το τόπο από το 10% προκειμένου να απελευθερωθούν τα επιπλέον 400 εκατομμύρια ευρώ το κάναμε με συνοπτική διαδικασία, πολύ γρήγορα και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί η πρόταση στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Και από ό,τι ξέρω και η Πολωνική Προεδρία δεν φύστη προσπαθειών προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία και να διεκπαιρεωθεί το θέμα τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και μάλιστα έχουμε συγκεκριμένα την ε, τροπολογία για να επιταχυνθούν τα μεγάλα ε, προγράμματα του Ταμείου Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε αυτή στην πρόκληση προκειμένου να ανακάμψει η ελληνική οικονομία. Φαντάζομαι και η ελληνική κυβέρνηση θα επιτείνει τι προσπάθειέ τη για να την αναθερμάνει. Γιατί αυτό που επιδιώκει η Ελλάδα είναι επαναφορά στον δρόμο τη ανάπτυξη και μάλιστα τη αηφόρου ανάπτυξη. Μια και δεν υπάρχουν άλλε ερωτήσει, ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ. Είστε πάντοτε ευπρόσδεκτο στην Επιτροπή μα. Ε, ιδιαίτερα όταν έχετε καλέ ειδήσει, Αυτέ μα ενδιαφέρουν περισσότερο, οι ειδήσει, αλλά Φυσικά και τα προβλήματα ε, που έχετε θα τα ακούσουμε ε, ευελπιστώντας ότι θα επιληθούν το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ. Meeting continues just if you give me two minutes. Δώστε απλώς δύο λεπτά να αποχαιρετήσω τον Υπουργό. Η συνεδρία συνεχίζεται. Dear colleagues, would you please... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε για να συνεχίσουμε. Dear colleagues, would you please take your seats? Yeah points Συνεχίζουμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι με το σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, τροποποίηση του κανονισμού 1083 του 2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένε διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική του σταθερότητα. Okay, as you Η πρόεδρος δεν επέστρεψε ακόμη. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας υποβάλει την πρόταση του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους σας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα βασικά σημεία, τους κύριους άξονες της πρώτης αναθεώρησης του κανονισμού 1083 για τον επιμερισμό του κινδύνου για τα κράτη-μέλη που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Οκτωβρίου. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μας κάλεσε για να παρουσιάσουμε σήμερα την πρόταση. Γιατί δεν είχαμε μέχρι στιγμής την ευκαιρία να εξετάσουμε την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο. Εξαιτία ε, της πληθώρας των συνεδριάσεων εκεί. Πριν περάσω στην ουσία της πρότασης, θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε δύο θέματα που κατά τη γνώμη μου έχουν κέρια σημασία ε, και διευκολύνουν και την περαιτέρω κατανόηση της πρότασης. Το πρώτο σημείο αφορά τη χρηματοδότηση ε, που σχετίζεται με δράση των διαρθρωτικών ταμείων και υπερβαίνει τις συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εθνική συγχρηματοδότηση. Και το δεύτερο σημείο αφορά τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις στις χώρες που μαστίζονται από την κρίση. Είναι γεγονός ότι η πολιτική της συνοχής προϋποθέτει στις περισσότερες χώρες σημαντικές, ε, σημαντικά ποσά συγχρηματοδότησης που προέρχονται είτε από τον ιδιωτικό είτε από το δημόσιο τομέα. Τέτοιου είδους χρηματοδότηση από τρίτο μέρος χρειάζεται στα πλαίσια των ε, σχεδίων που δημιουργούν έσοδα. Έχουμε το άρθρο 55 του κανονισμού που προβλέπει τους κανόνες ε, για την εφαρμογή σχεδίων που δημιουργούν έσοδα για το μέλλον. Εδώ όμως έχουμε μια προσέγγιση ε, με βάση του, του κενού που υπάρχει στη χρηματοδότηση σε σχέση με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και επιμερίζεται το επενδυτικό κόστος σε περίπτωση που δεν καλύπτεται αυτό από επιδοτήσεις των προγραμμάτων του Ταμείου Συνοχής. Ένα άλλο παράδειγμα αναφέρεται στις παραγωγικές επενδύσεις. Εκεί οι επενδυτές χρησιμοποιούν διάφορες πηγές χρηματοδότησης, ε, ακόμη και δάνεια ή επιδόματα, επιδόματα προκειμένου επιχορηγήσεις για να ε, δρομολογήσουν τέτοια προγράμματα. Σε κανονικές συνθήκες, οι δικαιούχοι των σχεδίων χρηματοδοτούν κόστος που δεν είναι επιλέξιμο για επιχορηγήσεις μέσω equity, equity δηλαδή ίδιους πόρους τις περισσότερες φορές ή μέσω χρέους, δανεισμού, είτε συνάπτοντας δάνεια είτε εκδίδοντας εταιρικά ομόλογα. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε και την εξή κατάσταση. Πολύ συχνά τα σχέδια χρηματοδοτούνται από μια επιχορηγήση, από ένα επίδομα ή κρατική ενίσχυση και ε, υπάρχει και συμπληρωματική ε, χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα. Έτσι λειτουργούν τα διαρθρωτικά ταμεία. Εμείς τώρα ασχολούμαστε με αυτό το τμήμα της ε, χρηματοδοτικής εισφοράς που υπερβαίνει όμως ε, το ποσοστό των επιχορηγήσεων που προέρχονται είτε από ευρωπαϊκές είτε από εθνικές πηγές. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχουμε με την κινητοποίηση ιδιωτικών κονδυλίων, ε, κονδυλίων από άλλες πηγές χρηματοδότησης είναι ακριβώ να χρηματοδοτήσουμε με αυτές τα σχέδιά μας, ιδιαίτερα στις χώρες που πλήττονται από την κρίση. Εκεί διαπιστώνουμε ότι οι ιδιωτικοί επενδυτές έχουν μειώσει δραστικά την έκθεσή τους σε κινδύνους, σε ανάληψη σχεδίου δηλαδή στη χώρα αυτή. Ακόμη και εθνικέ και κρατικέ τράπεζε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητα. Και η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα οξία στην Ελλάδα. Και μάλιστα ακούσαμε από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή σε πολλά μέτωπα. Και μάλιστα στην περίπτωση της Ελλάδας, ε, ένας μεγάλος αριθμός στρατηγικών και παραγωγικών επενδύσεων που καλύπτουν πολύ σημαντικά σχέδια στα πλαίσια των διευρωπαϊκών δικτύων, αυτή τη στιγμή διατρέχουν το κίνδυνο να μείνουν ανεφάρμοστα εξαιτίας της απροθυμίας των ιδιωτών επενδυτών που έχουν ενοχικές ε, υποχρεώσεις ε, συνδρομής στο πρόγραμμα ή εξαιτία άλλων περιορισμών των ε, διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών να παράσχουν περαιτέρω υποστήριξη σε τέτοιου του σχέδια. Και η κατάσταση αυτή επιταχύνεται εξαιτία της έλλειψη ρευστότητα από ε, ντόπιου επενδυτέ και από τις κρατικές τράπεζες. Στόχος της νέας πρότασης της αναθεώρησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπερβούμε το αδιέξοδο είναι η αναθεώρηση του κανονισμού και προτείνουμε ένα συνδυασμό των πόρων της ε, πολιτικής συνοχής με την δανειοδοτική ε, ικανότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε συνδυασμό με άλλα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα που έχουν κρατική λειτουργία, δημόσια λειτουργία παρόμοια με αυτή της ΕΤΕ. Τέτοιου χρηματοπιστωτικά όργανα μπορούν να συνεχίσουν να δανείζουν στις ε, χώρες που πλήττονται για να χρηματοδοτήσουν τα προγραμματά τους, συμπληρώνοντας τη χρηματοδότηση που απαιτείται προκειμένου να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή σχέδιο. Με βάση λοιπόν αυτό το ιστορικό θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ στο κυρίως ε, θέμα, στην αναθεώρηση του κανονισμού. Η πρόταση αναθεώρησης στηρίζεται σε υφιστάμενες διατάξεις του κανονισμού που προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, διαδραματίζει ειδικό ρόλο σε ό,τι αφορά, ιδιαίτερο ρόλο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των σχεδίων, ιδιαίτερα μεγαλεπίβολων σχεδίων και επίσης έχει ρόλο σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης και εταιρικών σχέσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο ιδιαίτερος ρόλος της ΕΤΕ που ήδη υπογραμμίζεται στον κανονισμό επισημαίνεται και στη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ε, Ευρωζώνης και των ε, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων που δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Στη δήλωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσκλήθηκαν να διευρύνουν τις συνέργειες μεταξύ των ε, διαφόρων προγραμμάτων και των κοινοτικών κονδυλίων στα κράτη-μέλη με διάφορους μηχανισμούς συνδρομής είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ε, Στι τρέχουσε συνθήκε όμω, η ΕΤΕ και άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί απαιτούν ε, επιπρόσθετες εγγύησεις προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν δανεισμό στις χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει στόχο να επιτρέψει ένα κράτος να ζητήσει συνδρομή από την Ένωση ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να χρησιμοποιήσει ένα τμήμα των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής προκειμένου να παράσχει εγγυήσει για δάνεια και άλλες χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις που στόχο έχουν την διευκόλυνση της εξασφάλισης χρηματοδότησης από τρίτο μέρος για τα προγράμματα αυτά και που αποτελούν τμήμα της στρατηγικής παρέμβασης της πολιτικής συνοχής στο δεδομένο κράτος μέλος. Αυτό που είναι σημαντικό να αντιληφθούμε είναι ότι έχουμε να κάνουμε μια σωρία προγραμμάτων που ε, σχετίζονται με την στρατηγική την πολιτική συνοχής, αλλά εστιαζόμαστε σε εκείνο το τμήμα των σχεδίων και προγραμμάτων που δεν την χάνει ε, ε Η πρόταση αυτή ανέκυψε μετά από τη συζήτηση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στοχεύει προς ε, να καλύψει στόχους και εγγύσεις ε, δάνει και εγγύη, συγγνώμη, της ΕΤΕ. Επίσης θέλει να μεγιστοποιήσει πιθανές ε, πηγές χρηματοδότησης με διετή ορίζοντα και επεκτείναμε την πρότασή μας προκειμένου να καλύψει και δεχόμενη ανάμειξη άλλων εθνικών ή διεθνών ε, δημοσίων φορέων που είναι σε θέση να παράσχουν παρόμοιες εγγύησεις με αυτές ε, της ομάδας ΕΤΕ. Για να δοθούν τέτοιες εγγύησεις δυνάμει των ε, κανόνων που ισχύουν για την επιμερισμένη διαχείριση, προϋποθέτει κάτι τέτοιο προποθέτει εκτενείς αλλαγές στον ε, κανονισμό του Συμβουλίου. Και ως εκ τούτου τροποποίηση και των εφαρμοστικών διατάξεων του κανονισμού. Με σημαντικές συνέπειες για την ομαλή εφαρμογή των διαφόρων μηχανισμών χρηματοοικονομικής τεχνικής που ήδη εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να μην προβούμε σε τέτοια ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση του εν λόγω κανονισμού. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι οι τεχνικές δυσκολίες που σχετίζονται με την προετοιμασία και τις διαπραγματεύσεις τέτοιου μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την περιορισμένη ε, θεσμική ικανότητα που έχουν τα μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την εφαρμογή τέτοιου μηχανισμού επιμερισμού κινδύνου μέσω ε, μίας έμεσης αλλά ε, κεντρικής διαχείρισης και όχι επιμερισμένης διαχείρισης. Κάτι τέτοιο συνάδει και με τις γενικές διατάξεις που χρηματοπιστω... του χρηματοπιστωτικού κανονισμού, του δημοσιονομικού συγγνώμη κανονισμού. Πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να χρησιμοποιήσει τα ισχύοντα μοντέλα μηχανισμών ε, επιμερισμού κινδύνου που ήδη εφαρμόζονται με βάση τον μηχανισμό έμεσης ε, επιμε, επιμερισμένης διαχείρισης και να χρησιμοποιήσει το, την κοινωτική χρηματοδότηση ως υπόδειγμα αυτό που κάνουμε για τις χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση ε, και την παροχή των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Τέτοιοι μηχανισμοί επιμερισμού κινδύνου εφαρμόζονται στα πλαίσια του 7ου ερευνητικού προγραμμάτος πλαισίου ή το ε, το μηχανισμό ε, εγγύησεων δανείων για διάφορα προγράμματα διασυνοριακά που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα και με πόρους των διευρωπαϊκών δικτύων. Αυτό το μοντέλο είναι το υπόδειγμά μας και αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό πάντως που πιστεύουμε είναι ότι Κατά τη γνώμη δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να προσδιορίσουμε με ακρίβεια όλους τους όρους και τις δυνατότητες ενός τέτοιου μηχανισμού επιμερισμού του κινδύνου. Στόχος μας είναι με την προτινόμενη αναθεώρηση του κανονισμού να συμπεριλάβουμε και μια ρήτρα που θα μας επιτρέψει να ελέγξουμε πιο διεξοδικά, να εξετάσουμε πιο διεξοδικά τη συγκεκριμένη αίτηση κράτους μέλους και να ανταποκριθούμε ανάλογα μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης. Στην αναθεώρηση αυτή δεν μπορούμε να είμαστε υπερβολικά διεξοδικοί και σχολαστικοί, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια διακριτική ευχαίρεια και κάποια ελαστικότητα. Επιπλέον, η χρηματοδότηση τέτοιων εργαλείων επιμερισμού του κινδύνου θα προέλθει αποκλειστικά από τους πόρους που ήδη έχουν κατανεμηθεί στα κράτη-μέλη δυνάμει των ισχυών των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. Ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει επιπρόσθετο βάρος για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τα χρήματα για την Ελλάδα, για παράδειγμα, θα προέλθουν από διατάξεις των ελληνικών προγραμμάτων και από κονδύλια που έχουν, μέχρι στιγμής δεν έχουν ε, προσδιοριστεί για συγκεκριμένα προγράμματα. Τέλος, αυτές οι, ε, οι συσφορές, αυτά τα κονδύλια που υπάρχουν και που θα δοθούν από τα κράτη-μέλη για τέτοιους μηχανισμούς επιμερισμού κινδύνου, θα πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά και να μην δημιουργήσουν προβλήματα στον κοινοτικό προϋπολογισμό ή ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή αυτής της αρχής. Επίσης υπάρχουν διατάξεις για την πιθανή επαναχρησιμοποίηση κάποιων κονδυλίων σε περίπτωση που μείνουν αναξιοποίητα κάποια κονδύλια και δεν καλύψουν συγκεκριμένες απώλειες, υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ε, επαναπροσδιορισμού των δαπανών. Βέβαια, θα πρέπει το κράτος μέλος να εξακολουθεί να είναι επιλέξιμο με βάση ένα πρόγραμμα συνδρομής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να γίνουν οι απαραίτητες μεταφορές σε περίπτωση που η συγκεκριμένη χώρα δεν είναι πια επιλέξιμη για το μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν είναι η βασική άξονα της πρώτες αναθεώρησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Sorry, I, I, I just... ε, λυπάμαι. Ε, θα ήθελα κι εγώ να πω το εξής. Ε, εγώ που είμαι αρμόδια για αυτή την έκθεση έχω καταλήξει στο εξής όπως λέτε και εσείς, ε, εδώ κατ' ουσίαν πρόκειται για μία ρήτρα που θα μας ε, επιτρέψει ε, να αναπτύξουμε ένα χρηματοψηφιακό εργαλείο το οποίο θα βοηθάσει να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εγώ σε γενικές γραμμές είμαι υπέρ αυτού του εργαλείου επιμερισμού κινδύνου όπως σε εποχές όπως τώρα όπου έχουμε χώρες που υποφέρουν πάρα πολύ από χαμηλή αξιολόγηση και από την έλλειψη ε, δανεισμού. Εδώ λοιπόν αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό όμως που με απασχολεί, εκεί που έχω επιφυλάξει, είναι διάφορα θέματα στον κανονισμό και θα τα συζητήσω αυτά με τους σκιώτες ηγητές ε, βέβαια εδώ πρόκειται για μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ε, μόλις ξεκινάει η διαδικασία. Νομίζω όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε τις χώρες εκείνες ε, που ε, μπορούν να είναι επιλέξιμες για ένα τέτοιο εργαλείο. Υπάρχει λοιπόν ένας ελάχιστος ε, κίνδυνος ε, ανασφάλειας στον τρόπο με τον οποίο ε, προσφέρουμε αυτή την ευκαιρία. Εδώ υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου θέλουμε να είμαστε περισσότερο ακριβείς. Και εγώ εξάλλου πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε με την Επιτροπή και με το Συμβούλιο κατά πόσον σε σχέση με αυτό το εργαλείο του επιμερισμού κινδύνου, κατά πόσον ε, αυτό θα πρέπει να γίνει ε, με διοικητική απόφαση ή ε, με διοικητική, διοικητική πράξη, εφαρμοστικό κανόνα μάλλον. Επειδή λοιπόν μόλις τώρα είμαστε στη φάση εισαγωγής αυτού του εργαλείου, είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι τα στοιχεία της περιφερειακής πολιτικής, ε, του συστήματος διαχείρισης, η Επιτροπή Ελέγχου, ε, πώς ορίζονται οι αποδέκτες, όλα αυτά που εντάσσονται μέσα στην πολιτική, που όμως δεν είναι απόλυτα σαφές ε, κατά πόσον ορίζονται ως σημαντικά στοιχεία για την δρομολόγηση αυτού του νέου εργαλείου. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά θεμάτων που έχουν σχέση με το πόσα χρήματα ε, μπορούν να ε, πρικοδοτήσουν αυτό το εργαλείο. Εδώ, όπως είπατε και εσείς, ε, απλά κάνουμε γενικές δηλώσεις. Δηλαδή, ανοίγει δυνατότητα να προβλεφθεί ένα τέτοιο εργαλείο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ, να δούμε τι μπορεί να ρυθμιστεί ποιοι είναι οι τομείς εκείνοι όπου πρέπει να υπάρξουν περισσότερες συζητήσεις. Και θα ήθελα να πω στους εσκιώδεις συζητητές μου ότι με ενημέρωσαν ποιοι είστε, ποιοι θα είστε, τα ονόματά σας. Ευχαριστώ τις πολιτικές ομάδες και αν κάποιος έχει προετοιμαστεί ε, να λάβει το λόγο σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πολύ ευχαριστώ να το κάνει, αλλιώς κάποια άλλη φορά. Ε, εσείς ε, με καλύψατε κατά το ίμιση. Αναφέρατε πολλά από τα πράγματα που ήθελα να πω. Θα ήθελα απλά να ζητήσω δύο διευκρινήσεις που έχουν σχέση με τις προτάσεις που ήδη ε, κατατέθηκαν. Πρόκειται για τη διαδικασία εφαρμογής για τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ποια θα είναι η διαδικασία, ε, ποιος είναι επιλέξιμος και ποιος ε, όχι. Νομίζω ότι αυτά είναι κάποια βασικά ερωτήματα. Και διαρωτώ με, όσον αφορά την τρίτη πρόταση, ε, κατά πόσο μπορούμε να μιλάμε για sunset clause. Και το άλλο που θέλω να μάθω είναι το χρονοδιάγραμμα, το timing αυτή της, αυτής της διαδικασίας. Ε, κατά πόσον θα σταματήσει ε, κατά την ε, αμέσως επόμενη περίοδο, υπάρχει κάποιο προηγούμενο. Αυτές είναι γενικές ερωτήσεις που είχα να κάνω, αλλά τα υπόλοιπα τα έφυξε έτσι κι αλλιώς συντανούτα και περιμένω τις απαντήσεις. Ο κύριος Βανίστερο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Πρόκειται για ένα καινούριο εργαλείο μέσο και αναφέρει ορισμένα στοιχεία που και εμείς τα ζητούσαμε πολύ καιρό. Το θέμα όμως είναι πρόκειται για κάτι θετικό, έτσι το κρίνει η Επιτροπή μας τουλάχιστον, αλλά παρόλα αυτά πρέπει στο επίπεδο του προϋπολογισμού να δούμε το θέμα με κριτικό πνεύμα. Δηλαδή, είναι όντως απαραίτητο να γίνουν αυτές οι αλλαγές με συμπληρωματικό τρόπο ή καλύτερα να το θέσουμε στα πλαίσια ενός καινούριου κανονισμού. Ίσως δεν είναι ο καταλληλότερος χρόνος εδώ, αλλά να τεθεί κάποτε. Ιβάν Γκουτμάν. Όχι, δεν είμαι ο ναι. Ιβάν. Εύερς λέγομαι, όχι Ιβάν. Καλά, με συγχωρείτε εμείς της Επιτροπής Προϋπολογισμού είπαμε ότι θα γράψουμε γνωμοδότηση και ότι μάλλον εγώ θα είμαι ο συντάκτης της και γι' αυτό ζήτησα το λόγο. Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Το 2009 πάνω από 6 δισεκατομμύρια χορηγήθηκαν ως πρόσθετες πληρωμές, τότε μπορεί να βοηθούσε αυτό. Αλλά για τις χώρες που έχουν πρόβλημα πάνω από 10% του ΑΕΠ τους ή που έχουν συμφωνία πληρωμών με την Κομισιόν χορηγήθηκαν άλλα διαφορετικά ποσά ως χρηματοδότηση. Τώρα λέμε να βοηθήσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα αρχής εδώ. Πρώτον, ποιον να βοηθήσουμε, διότι αν προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν πρόβλημα απορρόφησης, τότε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Οκτωβρίου, όχι δυστυχώς του Νοεμβρίου, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ ελλημάτων του προϋπολογισμού και ρυθμού απορρόφησης. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν μεγάλο πρόβλημα προϋπολογισμού, αλλά έχουν χαμηλό ρυθμό απορρόφησης. Το θέμα λοιπόν είναι με ποια κριτήρια, ποιες παραμέτρους θα εφαρμόσουμε για να επιλέξουμε τις χώρες που θα βοηθήσουμε. Γιατί αν δεν είναι συγκεκριμένα αυτά τα κριτήρια μπορεί να στοχεύσουμε λάθος. Και κάτι άλλο από απόψεως προϋπολογισμού που μπορεί να είναι επικίνδυνο. Αν η Τράπεζα Επενδύσεων δώσει εγγυήσεις στις τράπεζες των χωρών μελών ώστε να χορηγήσουν δάνεια για την αρχή της εφαρμογής ενός σχεδίου, τι θα γίνει άμα αποτύχει το σχέδιο. Ποιος τότε θα εγγυηθεί το δάνειο. Η Κομισιόν λέει ότι δεν είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό γιατί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για τη συνοχή είναι εγγυημένος. Αλλά αυτό είναι σαν το πρόβλημα της κότας και του αυγού. Το θέμα είναι ότι από την αρχή πρέπει να προβλέπετε αν θα δοθούν προκαταβολές και τι βαθμού και άρα Μπορεί αυτό να φαίνεται θετικό, αλλά από δημοσιονομικής απόψεως, αφού εμείς είμαστε αυτοί που ελέγχουν την ΕΤΕ, ποιος θα τη σώσει τις εγγυήσει που πρέπει να δώσει με τη σειρά της στις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θέλει κανείς άλλος να σχολιάσει. Α, ο Μάρκος Μπίμπερ. Ναι, ευχαριστώ. Άκουσα με προσοχή τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και έχω μεγάλες αμφιβολίες. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι όχι πολύ θετικό στην ουσία. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Συνοχής για να εγγυηθούμε νέες θέσεις για δάνεια σε ευρωπαϊκές τράπεζες, αν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις στον προϋπολογισμό για δάνεια, τότε συμφωνώ με αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής. Αν αποτύχουν τα προγράμματα, τι θα γίνει με τις εγγυήσεις τους. Εγώ έχω μεγάλες αμφιβολίες. Η κυρία Χιούμπνερ μίλησε για μία ρήτρα ενδυνάμωσης δυνατοτήτων. Ναι, αλλά όλα αυτά Ποιος θα τα ελέγχει, θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος, ποιος θα, έχει ποια δικαιοδοσία. Εγώ ως απλός βουλευτής ε, δεν καταλαβαίνω ακριβώς, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί κανείς να κρίνει το σύνολο της αξίας αυτής της πρότασης, ούτε πόσο χρόνος θα χρειαστεί για την εφαρμογή του. Είδα πόσο χρόνο χρειάστηκαν οι εκπρόσωποι της Κομισιόν για να υποβάλουν την πρόταση ενός μηχανισμού που πολλοί τον θεωρούν σαφή επιτέλους, αλλά πότε θα προλάβει το Κοινοβούλιο να τα εγκρίνει και να τα κρίνει όλα αυτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο εργαλείο για να ενισχύσουμε τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα έχουμε και πολλά ερωτηματικά και απορίες. Η πρόεδρος διακόπτη, γιατί δεν άκουσε τη διερμηνία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά και απορίες. Η συνοχή που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, πώς θα πραγματοποιηθεί. Αυτά τα κονδύλια, από πού θα προέλθουν, αυτή η τελευταία συγχρηματοδότηση. Γιατί υπάρχουν ορισμένες κυβερνήσεις που έχουν περισσότερα χρήματα και μεγαλύτερη ευρωστία, αλλά τι αποτέλεσμα θα έχει μια τέτοια κατάσταση στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό θα εχει μια τετοια κατασταση σε λιγοτερο ανεπτυγμενες χωρες αυτο θα πρεπει να το συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα για να δούμε αν η πρόταση αυτή και αν ο μηχανισμός που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως ευνοήσει μόνο τις ισχυρότερες κυβερνήσεις και τις ισχυρότερες χώρες, κάτι που αποβαίνει σε τελική ανάλυση εις βάρος της συνοχής, γιατί οι πιο αδύναμες χώρες έχουν περισσότερη ανάγκη υποστήριξη. Ο κύριος Τσέλερ. Äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε δεν μπορώ να υποβάλω τίποτε γραπτός. Άκουσα όσα υπόθηκαν, αλλά δεν μπόρεσα μέχρι τώρα να προετοιμαστώ κατάλληλα για αυτή τη συζήτηση. Ακούω ότι είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές και καταλαβαίνω ότι το, η πρόταση θέτει πολλά ερωτήματα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι Κάθε χρόνο το Δεκέμβριο όλες οι διοικήσεις ε, πυρετοδός ψάχνουν να βρουν τα, πώς θα καλύψουν τα ελλείμματα στον προπολογισμό τους. Αλλά ο σκοπός είναι να τον προετοιμάζετε τον προπολογισμό σας καταλήλως ώστε να μην χρειάζονται τέτοιου είδους επίγοντα μέτρα κάθε τέλος, κάθε χρόνο. Έχω ακούσει ότι παρόμοιες δαπάνες ε, σχεδιάζονται και αλλού. Και θα ζητηθεί λέει από την Ετένα της χρηματοδοτήσει. Άρα να χρησιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ελλείψεις των προϋπολογισμών, αλλά η ΕΤΕ δάνεια κάνει και μάλιστα όχι δωρεάν. Εμάς θα μας κοστίσει κάτι αυτό. Εάν δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια, θα χρειάζονται συνεχώς δανεισμοί και θα αυξάνουν τα επιτόκια. Δεν μου φαίνεται πολύ σωστή ιδέα. Πρέπει να υπολογίσουμε, να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι ότι λέγω δεν υπάρχουν πάντα και για, όλα δυνατότητες συγχρηματοδότησης. Πώς θα πληρώσουν, θα αποπληρώσουν τα χρέη τους οι χώρες που θα έχουν λάβει τέτοιου είδους δάνεια της ΕΤΕ αν δεν μπορούν ήδη από τώρα να συγχρηματοδοτήσουν. Ή μήπω αυτό θα αποτελέσει ευκαιρία μόνο για όσους έχουν κάποια χρήματα, αλλά δεν μπορούν, δεν είναι αρκετά για να τα συγχρηματοδοτήσουν αυτά τα προγράμματα. Δεν είναι σαφή τα πράγματα. Ούτε ήταν αυτός ο στόχος, ο αρχικός στόχος του προγράμματος. Ήταν να βοηθήσει τις περιφέρειες και χώρες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δεν θέλουμε να τις ενθαρρύνουμε τις περιφέρειες αυτές και τις χώρες αυτές να πάρουν περισσότερα δάνεια, αλλά να αναπτυχθούν πιο σοβαρά στο μέλλον. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ξαναδούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και με γραπτό τρόπο για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε και εμείς γραπτά. Η κυρία Ματσόνη. Ευχαριστώ. Εστερνίζομαι και εγώ τον προβληματισμό και τις απορίες των συναδέλφων. Θα ήθελα να προσθέσω μία ερώτηση διαδικαστική. Φαντάζομαι ότι αυτή η αναθεώρηση θα περάσει με τη συνοπτική διαδικασία, όπως ίσχυσε και για την προηγούμενη αναθεώρηση, που θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Ή όχι. Όχι. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων, Κλαρίσα. Αυτό αφορούσε τι προηγούμενε τροπολογίε. Τώρα περάμε στην τρίτη αναθεώρηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ναι, αλλά η ερώτησή μου είναι, θα έχουμε και πάλι το... τη συνοπτική διαδικασία γιατί... που ίσχυσε και την προηγούμενη αναθεώρηση του 1983 θα είναι τόσο πιεστικό το χρονοδιάγραμμα όπως και προηγουμένως, γιατί είναι πολλά τα θέματα και ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για την εξέτασή τους. Ερωτώ επίσης αν τα, τα, τα κονδύλια που αναφέρονται είναι τα κονδύλια των προηγούμενων χρόνων, δηλαδή αχρησιμοποιητή κονδύλια από το σύνολο του προγραμματισμού του, του προϋπολογισμού που αφιερώνεται σε συγκεκριμένη χώρα. Αυτή τη διευκρίνηση θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ποια χρησιμοποιεί τα κονδύλια, αναφέρεται ο Φρανσουά Αλφονζή. Αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό της επιφυλάξης και της απορίες των συναδέλφων, αλλά μην ξεχνάτε ότι η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη, ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου που μαστίζονται πιο πολύ από την κρίση. Και αυτό το μέτρο στόχο έχει να επιβλέξει κάπως την κατάσταση και να στηρίξει τις ε, προσπάθειες εξηγήσεις που κάνουν οι χώρες αυτές. Οπότε μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να την εξετάσουμε όχι με σκεπτικισμό και επιφυλακτικότητα, αλλά με πνεύμα συνεργασίας προς τις χώρες του Νότου. Mm. Γιατί στο μέλλον δεν θα μιλάμε πια μόνο για ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Θα πρέπει να ατενίζουμε και το μέλλον και να υιοθετήσουμε πιο επικοδομητικά σχέδια για τις χώρες που σήμερα μαστίζονται από την κρίση. Η Πρόεδρος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση και να πω και εκ μέρους των σχεδόν εισηγητών ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων, γιατί με τις απορίες φάνηκα τα σημεία που χρήζουν διευκρίνησης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να απαντήσει όσες ερωτήσεις μπορεί και επίσης να σας ενημερώσω ότι όταν ο Διευθυντής Νίσλερ θα ολοκληρώσει την παρουσίασή του, δεν χρειάζεται να λάβουμε σήμερα κάποια απόφαση, γιατί σήμερα είναι η απαρχή της συζήτηση και δεν ισχύει η συνοπτική διαδικασία fast track για τη συγκεκριμένη τρίτη τροπολογία, όπως ίσχυε για τις προηγούμενες δύο. Σε πέντε λεπτά θα πρέπει να πάω σε άλλη συνεδρίαση για να παρουσιάσω την πολιτική μου. Θα αφήσω στο πόδι μου τον Γιώργο Σταυρακάκη μετά την παρουσίαση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ρούντολφ Νίσλερ, θα περάσουμε στην επόμενη, στο επόμενο θέμα της σας διάταξης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χιούμπνερ. Θα ήθελα στη φάση αυτή να πω ότι περίμενα, α, φανταζόμουν ότι θα υποβάλλετε τόσες ερωτήσεις, γιατί όντως η πρόταση που καταθέσαμε mm-hmm. είναι μια πρόταση που υπερβαίνει κάπως το, το ρόλο και τους τομείς που καλύπτει η πολιτική συνοχή. Είναι μια πρόταση που δίνει τη δυνατότητα δημιουργία νέων μηχανισμών και εργαλείων προκειμένου κάποια κονδύλια να περνάνε την πολιτική συνοχή στο σύστημα άμεσης διαχείρισης. Αυτό λαμβάνει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΤΕ που είναι εταίρος της και εφαρμόζεται με βάση τους γενικούς κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτό είναι κάτι που πρώτη φορά συζητούμε στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλές απορίες. Πάντως πολύ ευχαρίστω ε, με το επιτελείο μου να σας διαλευκάνουμε όλα τα επιμέρους στοιχεία αυτής της πρότασης για να λυθούν οι απορίες σας. Κύριε Αλφόνση, ε, όπως είπατε, αυτό το μέτρο είναι συμπληρωματικό προκειμένου να στηρίξει το, την εφαρμογή άλλων μέτρων της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι ο στόχος της αναθεώρησης. Τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο. Θέλουμε να βρούμε ένα τμήμα χρηματοδότηση που δεν καλύπτεται από τους κανόνες της πολιτικής συνοχής. Δηλαδή δεν πρόκειται ούτε για κοινοτική συνεισφορά, ούτε για νοσιακή συνεισφορά, ούτε για συγχρηματοδότηση εθνική. Αυτά τα θέματα τα καλύψαμε αλλού στην πρόταση, προκειμένου να βοηθήσουμε μιας χώρες, μία, να βοηθήσουμε τις χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση μέσω του top-up. Εδώ έχουμε ένα πλέον τμήμα που συνήθως συνδέεται με τη στρατηγική και τα σχέδια της πολιτικής συνοχής αλλά εκπίπτει κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση. Αλλά είναι απαραίτητο και το τμήμα αυτό για να εφαρμοστούν επιπλέον τα, τα προγράμματα. Ε, οι παραχωρήσει των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων είναι ένα μεγαλεπίβολο έργο πολλών δισεκατομμυρίων και πάνω από το μισό τη χρηματοδότηση προέρχεται από πηγέ που δεν είναι ούτε ευρωπαϊκές ούτε εθνικές. Είναι ε, συνεισφορές του ιδιωτικού τομέα και αυτές οι συνεισφορές λείπουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και έχουν ε, κινητοποιηθεί οι διαδικασίες αυτές ε, για τις παραχωρήσεις των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων. Θέλουμε να επιβλέξουμε την κατάσταση, να ε, συνεχίσει η ροή των ιδιωτικών κονδυλίων για, να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα από τις ελληνικές αρχές. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα, ποιο, ποια χώρα είναι επιλέξιμη. Σίγουρα το ελληνικό παράδειγμα μας ενέπνευσε μας ενέπνευσε έγινε μια διεξοδική ανάλυση αυτού του φαινομένου και αυτής της κατάστασης και είπαμε ότι ε, βρισκόμαστε σε, μια, σε ένα πλαίσιο δρυμύτατης κρίσης, όπως σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και βέβαια μπορεί να ισχύει και για άλλες χώρες που τη χάνουν στήριξη είτε από κοινοτικό πρόγραμμα, μηχανισμό στήριξη είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτές είναι οι επιλέξιμες χώρες που έχουν έλλειψη ρευστότητας και δεν ε, καλύπτονται, δεν ικανοποιούνται ούτε από το top-up. Υπάρχει τώρα μία διαφορά σε ό,τι ε, αφορά το κατά πόσο μπορούμε με αποτελεσματικό τρόπο να εφαρμόσουμε τέτοια μέτρα στήριξης. Γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει διεξοδικότατη ανάλυση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία περιπτωσιολογική ανάλυση. Αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα ισχύσει αυτή αυτό το μέτρο, αυτός ο μηχανισμός για όλες τις χώρες που πλήττονται από την κρίση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρετε θα γίνει μια περιπτωσιολογική ανάλυση και είναι και σημαντική διαφορά σχέση με τις προηγούμενες μας προτάσεις. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να γίνει κατανοητό το επισήμανε ο κύριος Πίπε. Που είναι το τελευταίο βιολί κατά κάποιο τρόπο, όπως λέμε. Δηλαδή, δεν είναι να ξοδέψουμε χρήματα που έμειναν στο τέλος του έτους ανεκμετάλλευτα. Στόχος μας είναι να ξεμπλέξουμε την κατάσταση σε ορισμένα προγράμματα που χρήζουν ε, ιδιωτικής συνεισφοράς. Γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε τη συγκεκριμένη θεώρηση για να επαναφέρουμε τη ροή των ιδιωτικών κονδύλιων. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πώς θα συνδυαστούν αυτοί οι κανόνες με την πολιτική συνοχή και, τους, και τις γενικές διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, μην ανησυχείτε, έχουμε δύο μηχανισμούς, το LGTT και το RSFF. Αυτά τα δύο εργαλεία εφαρμόζονται με βάση τις διατάξεις που θα εφαρμόσουμε και εδώ και υπάγονται στον πλήρη έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εφαρμόζονται από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με ενοχικές συμφωνίες ε, συμβατικές που έχουμε. Δεν είναι κάτι που θα ξεκινήσει εκ του μηδενός δηλαδή. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους δύο μηχανισμούς και αυτή την εμπειρία και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι εν ευθέτω χρόνο. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπα πάντως, είμαστε στη διάθεσή σας για να δώσουμε περαιτέρω εξηγήσεις και πληροφορίες για να γίνει αντιληπτή η πρότασή μας. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας και τώρα πάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα ξεκινήσει η συζήτηση για το σύνολο των κανονισμών και προτείνω το εξή. Ο Γενικό Διευθυντής, ο κ. Νικόλα Μαρτίν, θα κάνει την εισηγησή του, μετά οι εισηγητέ και αν υπάρχει χρόνος θα δώσουμε και ε, χρόνο στου και γιατί όπω ξέρετε να τελειώσουμε σε έξι. Παρακαλώ, ε, έχετε το λόγο. Ο κ. Νικόλα Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να έρθω εδώ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης που μου δίνεται η δυνατότητα μετά την έγκριση της, των προτάσεων για το ρυθμιστικό πακέτο, την έγκριση από την Κομισιόν, ευχαριστώ που μπορώ να σας παρουσιάσω αυτό το θέμα εδώ. Ε, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Από την άλλη βέβαια έχουμε και ένα αρκετά περίπλοκο πακέτο κανονισμών. Εκείνο το οποίο θα κάνω είναι να δράξω την ευκαιρία για να σας παρουσιάσω σύντομα μια γενική επισκόπηση των βασικών στοιχείων του πακέτου που θα αποτελέσουν τη βάση για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Βεβαίως ε, είμαι στη διάθεσή σας ε, για να εμβαθύνουμε σε κάποια στοιχεία. Νομίζω λοιπόν ότι το άτυπο έγγραφο εργασίας το οποίο προετοίμασε ο εισηγητής για τον κανονισμό κοινών ε, διατάξεων, αυτό αποτελεί μια πολύ καλή βάση γιατί προβάλλει βασικά στοιχεία της πρότασης της ε, Κομισιόν και καταδεικνύει ορισμένα από τα θέματα τα οποία πράγματι χρήζουν ε, εντελεχούς εξέτασης. Το πακέτο, όπως είπαμε, είναι αρκετά περίπλοκο, διότι ε, περιλαμβάνει ε, ένα γενικό κανονισμό ε, που έχει κοινέ διατάξεις και δεν αφορούν μόνο τα ταμεία συνοχής, αλλά αφορούν και την γεωργική ανάπτυξη και την αλία. Και μετά έχουμε πολύ συγκεκριμένου κανονισμού ε, που αφορούν το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη, συνοχή το Κοινωνικό Ταμείο ε, και έναν ξεχωριστό κανονισμό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Επίσης έχουμε και έναν ε, άλλο κανονισμό για το EGTC. Όλα αυτά αποτελούν το πακέτο μας. Εγώ λοιπόν θα ασχοληθώ περισσότερο με το γενικό κανονισμό και μετά θα πω λίγα λόγια για τον ε, συγκεκριμένο κανονισμό του Ταμείου, όχι για τον ε, κανονισμό EFSF, ο οποίος ε, θα παρουσιαστεί στην αρμόδια επιτροπή. Είναι λοιπόν σωστό νομίζω να υπογραμμίσουμε ότι οι στόχοι που αναφέρονται για την πολιτική συνοχή, οι στόχοι αυτοί έχουν κάποια συνέχεια με την έννοια ότι προσφέρουν τη συνέχεια με το άρθρο 174 της συνθήκης. Αυτό βέβαια είναι κάτι που υπογραμμίζει τις προτάσεις Κομισιόν και ε, προσφέρει και τον σύνδεσμο με την στρατηγική της Ευρώπης 2020. Μία από τις άλλες αλλαγές είναι ότι προβλέπουμε δύο στόχους αντί των στόχων που ξέρετε από παλαιότερες ε, περιόδους το στόχο της ε, σύγκλησης, το στόχο της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε λοιπόν δύο στόχους ε, επενδύσεις για ανάπτυξη ε, και ε, θέσεις εργασίας και την ευρωπαϊκή περιφερειακή συνεργασία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πολιτική είναι πολιτική επενδύσεων για όλες τις περιφέρειες και υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά στο επίπεδο χρηματοδότησης των διαφόρων περιοδοχών. Θα προχωρήσω γρήγορα. Ε, μπορείτε μετά να δείτε και τις ε, διαφάνειες. Ε, κάποια, κάποιες διαφάνειες περιλαμβάνουν και στοιχεία αναφοράς. Φαντάζομαι θα γνωρίζετε και πώς ακριβώς γίνεται η κατανομή σε δύο-τρεις κατηγορίες περιφερειών. Και περιλαμβάνονται και κάποια άλλα στοιχεία από την πρόταση της Κομισιόν που συμπεριλήφθηκαν και στην πρόταση MMF ένας νέος κανονισμός ο οποίος ε, αφορά ε, τόσο την, ε, το phasing out το περίφημο, αλλά και άλλες περιοχές. Εκείνο λοιπόν το οποίο προβλέπεται για ειδική μεταχείριση είναι ένα δίκτυο ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι πράγματι υπάρχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο χρηματοδότησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία μετάβασης. Ε, και εδώ ε, βλέπετε πάλι μία διαφάνεια που χρησιμεύει για αναφορά. Έχουμε διάφορες κατηγορίες ε, περιοχών με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, αλλά βεβαίως είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι τα τελευταία στοιχεία του ΑΕΠ χρησιμοποιούνται για τον τελικό ορισμό των περιοχών. Και εδώ ε, θα ήθελα να φέρω λίγα λόγια για το Ταμείο Συνοχής. Βλέπετε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη που ε, ενδείκνυνται ε, για το Ταμείο Συνοχής. Αυτό με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και την προσέγγιση που υπάρχει ε, σε σχέση με τις ε, επενδύσεις στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μπορούμε λοιπόν να δούμε λιγάκι τον τρόπο με τον οποίο ε, θα ενισχυθεί το στρατηγικό, ο στρατηγικός σχεδιασμός. Νομίζω ότι αυτό υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούμε να ενισχύσουμε ε, την συνεργασία και την διαχείριση σε, σε πολλά επίπεδα. Βλέπετε λοιπόν την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μέσα από την εισαγωγή ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Συμπεριφοράς. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η έκθεση της Κομισιόν, ε, το οποίο στοιχείο αποτελεί σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της αρχής της συνεργασίας και αυτό μέσα από ένα κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος ε, μπορεί να εγκριθεί μέσα από κατεξουσιοδότηση πράξη. Και ε, έτσι λοιπόν αυτό για να διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά η συνεργασία και ότι υπάρχουν ε, διάφοροι τρόποι επιτυχίας, επίτευξης μάλλον της πολλαπλούς διακυβέρνησης. Επίσης έχουμε και άλλα βασικά στοιχεία που αναφέρονται στις κοινέ διατάξεις και έχουν σχέση κυρίως με την ισότητα των φύλων, τη μη διακριτική μεταχείριση και την προαγωγή της αηφόρου ανάπτυξης. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο στοιχείο της στρατηγικής προσέγγισης, που είναι η διασύνδεση με την στρατηγική του 2020. Για να επιτύχουμε το στόχο μας, πρέπει να έχουμε ένα κατάλογο θεματικών προσεγγίσεων που προέρχονται από αυτή τη στρατηγική του 2020, ε, αυτά βεβαίως ε, ε, αφορούν και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες για να καλυφθούν οι 11 βασικές περιοχές για επενδύσεις. Αυτό που παίζει επίσης ρόλο είναι ότι αυτά αφορούν και τα πέντε ταμεία, αφορούν το σημείο αναφοράς και τα ταμεία τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Υπάρχει τώρα και ένας μηχανισμός για να μεταφέρουμε όλα αυτά σε συγκεκριμένο προγραμματισμό. Ξεκινάμε με το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Είναι το έγγραφο το οποίο προβλέπεται ότι θα εγκριθεί από την Επιτροπή και εκεί θα αναφέρεται μία ολοκληρωμένη στρατηγική επενδύσεων των ταμείων. Και έτσι τα κονδύλια θα χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για να επιτευχθούν οι στόχοι. Μιλάμε για ένα σημείο αναφοράς του σχεδιασμού που θα γίνει στα κράτη-μέλη. Ξεκινάμε με τους ε, θεματικούς στόχους, πάμε πιο κάτω στις ε, προτεραιότητες και μετά εντοπίζουμε τους ε, τομείς τους οποίους πρέπει να γίνουν επενδύσεις και προσφέρονται και οδηγίες για το πώς θα γίνεται ο συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και πώς θα γίνεται και η διασύνδεση ανάμεσα στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τους συγκεκριμένους στόχους. Ε, κατόπιν, σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιείται το CSF, ε, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, ω σημείο αναφοράς. Ένα, μία σύμβαση συνεργασίας ανακράτος ε, μέλος, αλλά με αυξημένη συνεργασία και πιο δυναμικές ιδιότητες. Αυτά όταν σε ένα κράτος μέλος υπάρχει αποκριστάλλωση των συζητήσεων έτσι ώστε να γίνουν οι τελικές επιλογές που θα διοχετευτούν τα, διοχετευτούν τα κονδύλια ε, και ε, το ε, σχέδιο το εταιρικό τα καλύπτει όλα αυτά και παρουσιάζεται στην Κομισιόν για να γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Μιλάμε για ένα και μόνο έγγραφο ανακράτος μέλος, το οποίο ε, κάνει μία σύνθεση ε, του πώς θα χρησιμοποιούν τα κονδύλια, γίνεται διαχωρισμός σε διάφορους ε, θεματικούς στόχους. Όλα αυτά διασυνδέονται με την περιφερειακή στρατηγική, η οποία έχει ως στόχο να προβάλλει την χρήση, τις επιλογές που γίνονται. που παίζει ρόλο είναι να διασφαλίσουμε το συντονισμό και την αποτελεσματική εφαρμογή. Πέρα από αυτό και δεν έχω σχετική διαφάνεια, έχουμε και εφαρμοστικά προγράμματα που θα τα ξέρετε βέβαια, Αυτά όμως ε, περιλαμβάνουν και λεπτομέρειες ε, όσον αφορά στην επιλογή των προτεραιοτήτων. Εγώ θα εστιάσω την προσοχή μου σε ορισμένα νέα ε, στοιχεία. Ε, όλα τα άλλα αφορούν στο πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ε, της ε, πολιτικής, της πολιτικής συνοχής. Υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί που προβλέπουν κάτι τέτοιο και ορισμένοι εξ αυτών προσφέρουν και την επιλεξιμότητα. Υπάρχει επιλεξιμότητα εξάντε για να αποδείξουμε ότι πριν αρχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα ισχύουν κάποιες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για να επιτύχουμε την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Υπάρχει λοιπόν ένα παράρτημα στον κανονισμό που για την πολιτική συνοχής για κάθε θεματική προσέγγιση αναφέρει βασικούς στόχους, στρατηγικές και αυτά είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση αυτοαξιολόγηση από το κράτος μέλος, μετά ακολουθεί εξέταση από την Κομισιόν και αν δεν υφίστανται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε σε σοβαρές περιπτώσεις δεν θα ξεκινήσει η ροή των κονδυλίων. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να έχει διασφαλιστεί ότι είναι έτοιμο το έδαφος για την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Πάμε τώρα σε μία δεύτερη μορφή επιλεξιμότητας. Είναι η γνωστή μακροοικονομική επιλεξιμότητα που συνδέει την πολιτική συνοχής με την... Ε, ε, ναι. Στην περίπτωση των κρατών μελών, οι προϋποθέσεις ε, ορίζονται Υπάρχει λοιπόν ένας τρόπος με τον οποίο η Κομισιόν μπορεί να ζητήσει αλλαγές ε, στα προγράμματα έτσι ώστε τα κονδύλια να αναδιοχετεύονται ε, και να υπάρχει η βέλτιστη δυνατή χρήση για να στηρίζονται οι προτάσεις του Συμβουλίου. Όταν ένα κράτος μέλος δεν έχει εφαρμόσει σωστά τις συστάσεις ε, του Συμβουλίου ή αν δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να λάβει οικονομική βοήθεια, τότε υπάρχουν διατάξεις για την αναστολή των πληρωμών. Στην ε, τρίτη μορφή της ε, αιρεσιμότητας πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα διοχετεύονται για την επίτευξη των στόχων. Η ιδέα είναι η Για κάθε πρόγραμμα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο εντοπίζει τα ορόσημα και αυτά σχετίζονται κατόπιν με την επίτευξη των στόχων, με μία σειρά δικτών, ε, με το αποτέλεσμα και την απόδοση. Και έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε ένα μηχανισμό παρακολούθησης που σημαίνει ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει απολογισμός για το κατά πόσον οι ενός προγράμματος είναι σωστές ή όχι. Αυτό που παίζει επίσης ρόλο είναι να δούμε ε, κατά πόσον η προτεραιότητα συνδέεται και με την απόδοση. Για κάθε κράτος μέλος υπάρχει ένα αποθεματικό ε, της ε, απόδοσης programs uh, on the basis of the assessment made in Ιδιαίτερα στα πλαίσια των, της αξιολόγησης που έγινε στη στρατηγική του 2020. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις και εκεί υπάρχουν δυνατότητες αναστολής. Ε, μπορεί να γίνουν και ε, διορθώσεις σε ένα πρόγραμμα. Θα ήθελα τώρα να επισημάνω σύντομα και ένα-δύο άλλα στοιχεία ε, που αφορούν στην ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κοινοί κανόνες για όλα τα ταμεία. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε ε, μία ε, θεώρηση ε, από κάτω προς τα πάνω είναι μία χρήσιμη προσέγγιση για να επιτύχουμε ένα συγκεκριμένο είδος τοπικής ανάπτυξης. Αυτοί είναι κανόνες που βοηθούν όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία να βελτιώσουν τη στρατηγική τους και να εφαρμόσουν τη χρηματοδότηση με συντονισμένο τρόπο. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, μάλλον τα εργαλεία χρηματοδότησης, έχουμε μάθει πάρα πολλά ε, για τη χρήση τους ε, και μάθαμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο ε, το οποίο θα έρει περιορισμούς και θα διασφαλίζει ότι ευθύς εξ αρχής υπάρχουν σαφείς κανόνες. Θα χρησιμοποιείται η εμπειρία για να δοκιμαστούν οι ρυθμίσεις αλλά και για να εισαχθούν και νέες συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να υπάρχει χρήση πλατφόρμας χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και ειδικά κονδύλια ε, για τα οποία θα υπάρχει και η εγγύηση ότι είναι απόλυτα συμβατά αυτό, αυτά θα είναι ε, standard μοντέλα τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν ε, τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία ολόκληρη σειρά επιλογών που μπορούν να διευκολύνουν τη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Εδώ πολύ δύσκολα, ε, πολύ γρήγορα με θέλω να επισημάνω ένα από τα επιτεύγματα των προτάσεων. Δηλαδή υπάρχουν κοινοί κανόνες που διέπουν την αιρεσιμότητα των κονδυλίων Έχουμε μάθει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη ε, να χρησιμοποιούν το απλουστευμένο κόστος. Αυτό το μοντέλο. Και νομίζω αυτό το μοντέλο πρέπει να το ε, διαδώσουμε και να θέσουμε σε ισχύ τις ε, σχετικές διατάξεις για να είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Τέλος, θα ήθελα πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω τις ρυθμίσεις χρηματοδοτικής διαχείρισης. Εδώ πολλά συνδέονται με την πρόταση της Κομισιόν για την αναθεώρηση του ε, ε, χρηματοδοτικού κανονισμού. Αυτά τα έχουμε εντάξει και στην πολιτική συνοχή. Έχουμε μία ε, διαδικασία πιστοποίησης που είναι αυτή καινούργια, ένα κράτος μέλος ορίζει έναν ε, τομέα φορέα πιστοποίησης, ε, ο οποίος ορίζει κατόπιν και τον φορέα διαχείρισης. Δηλαδή, ε, η λογοδοσία πάει από το κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιορίζομαι την συμμετοχή της Κομισιόν στην όλη διαδικασία. Εξάλλου σε αιτήσια βάση έχουμε εκαθάριση λογαριασμών ε, με βάση τις δηλώσεις που γίνονται ε, και υπάρχουν και κάποια νέα στοιχεία ε, τα οποία προβλέπουν το ετήσιο κλείσιμο έτσι ώστε η έλεγχη να είναι περισσότερο αναλογική. Αυτές τις μεθόδους επιλέξαμε για να πλουστεύσουμε το σύστημα. Αλλά και πάλι σας λέω ότι τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να μπούμε σε λεπτομέρειες. Τώρα πάω σε άλλο θέμα. Ε, μία γενική επισκόπηση ε, των ε, κανονισμών που αφορούν τα κονδύλια. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί που προβλέπονται, καινούργοι, ιδιαίτερα ως προς τη στήριξη τομέων που καλύπτονται από το πρόγραμμα συναλλαγών εκπομπών, παραγωγής καπνού, πυρηνικών σταθμών και άλλων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Και υπάρχουν επίσης περιορισμοί και στη στήριξη μεγάλων, ιδιαίτερα μεγάλων επιχειρήσεων. Υπάρχει δηλαδή πιο συγκεκριμένη στόχευση και δεν χορηγούνται όλα αυτά τα κονδύλια γενικά για παραγωγικές επενδύσεις. Επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες ε, προβλέψεις για το θέμα της συγκέντρωσης των επενδύσεων σε προκαθορισμένες επιλογές, προτεραιότητες. Παραδείγματος χάρη η κίνηση προς οικονομία με χαμηλότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Βλέπουμε ότι έχει προταθεί ένας νέος μηχανισμός όπου υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ μεταβατικών και περισσότερο αναπτυξιακών προγραμμάτων από τη μία και λιγότερο ανεπτυγμένων ή αναπτυξιακών προγραμμάτων από την άλλη και μάλιστα με τρεις συγκεκριμένους θεματικούς στόχους που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες, την αποτελεσματική χρήση, η αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, ανταγωνιστικότητα και, και λέγω την καινοτομία ανανεώσιμες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα λοιπά αυτά που είπα. Βλέπετε εδώ τα ποσοστά στη διαφάνεια τουλάχιστον 20% πρέπει να διατεθεί στην αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες προβλέπουμε 50% της χρηματοδότησης να χρησιμοποιηθεί για αυτούς τους τρεις θεματικούς στόχους 6% τη χρηματοδότησης για τις ανανεώσιμες και τις, την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας στις αν λιγότερο αναπτυγμένες επαναλαμβάνω περιφέρειες. Θα ήθελα να σας ξαναπώ ότι να ξανατονίσω τον τρόπο με τον οποίο προβλέπουμε το μηχανισμό περισσότερης ορατότητας επενδύσεων σε αστυνομία κά προγράμματα τουλάχιστον 5% δηλαδή των πόρων μας να χρησιμοποιούνται για αστική ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βιώσιμη μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν έχω όσο χρόνο θα ήθελα, αλλά είναι σημαντικό να τονίσω τα γενικότερα στοιχεία του κανονισμού. Θα συντομεύσω γιατί το υπόλοιπο της παρουσίασής μου αφορούσε πιο λεπτομερή θέματα και ας περιοριστώ όμως τα σημαντικότερα άσα. Άρα σταματώ εδώ. Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ Διευθυντά για την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Κατάλαβα ότι υπήρξε μια παρεξήγηση. Είχα πει ότι ο λόγος θα δοθεί πρώτα στους εισηγητές για όλους τους κανονισμούς και μετά στους σκιώδεις αν υπάρχει χρόνος. Αρχίζω λοιπόν, αρχίζω λοιπόν με την Κωνσταντζα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το να πιστεύετε ότι σε μισή ώρα μπορούμε να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική για το νομοθετικό πακέτο και την πολιτική συνοχής. Βέβαια κανείς ε, δεν φταίει γι' αυτό και σίγουρα όχι ο κύριος Μάρτιν. Εγώ όμως προτείνω αύριο να αλλάξουμε την ημερησία διάταξη, να διαγράψουμε τα σημεία 12 και 13, να μην τα συζητήσουμε και να συνεχίσουμε με αυτό το θέμα αύριο το πρωί. Γιατί για τους εισηγητέ είναι σημαντικό ε, πριν καταλήξουμε σε έγγραφο εργασία, να γίνει πρώτα σοβαρή κουβέντα εδώ στην Επιτροπή. Ε, η δουλειά είναι αρκετά δύσκολη. Ε, και νομίζω ότι οι εισηγητές μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν, ωραία πράγματα, αλλά αν από την αρχή δεν προσπαθούμε να βρούμε εδώ στην Επιτροπή μας τη συνένεση, ποτέ δεν θα υπάρξει συνένεση και σίγουρα όχι τέλος του 2012. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ θερμότατα η συζήτηση να συνεχίσει και αύριο το πρωί. Επιτρέψτε μου τώρα να ξεκινήσω και θα αρχίσω να μιλάω για τον γενικό κανονισμό. Εσείς μας παρουσιάσετε ένα πρώτο έγγραφο εργασίας και εγώ θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα να σας παρουσιάσω ε, τα θέματα που με ενδιαφέρουν. Αλλά κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε χρόνο και αν θέλετε τον Ιανουάριο να προβλεφθεί μια ειδική συνεδρία της Επιτροπής όπου θα ασχοληθούμε μόνο με αυτό το πακέτο. Δεν είναι δυνατόν το πακέτο αυτό να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας κανονικής συνεδρίασης. Και αυτό τη στιγμή μάλιστα που οι προκλήσεις είναι πολλές. Εκείνο το οποίο χαιρετίζω είναι ότι η Κομισιόν με αυτόν τον κοινωνικό κανονισμό κατέθεσε μία πρόταση όπου δεν περιλαμβάνεται μόνο η πολιτική σύνοχης αλλά και η πολιτική γεωργία, το Γεωργικό Ταμείο και το Ταμείο Αλίας. Mm. Μιλάμε για έναν κανονισμό ομπρέλα ο οποίος ο κανονισμός ε, θα συμβάλλει στην απλούστευση των διαδικασιών. Και χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός αυτό. Μόνο που αυτό σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να επιδείξουμε τεράστια πειθαρχία στη δουλειά μας και στη συνεργασία με άλλες επιτροπές. Αυτό δεν είναι εύκολο και να οργανωθεί μάλιστα. Κατόπιν τούτου πρέπει να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που υπάρχει ε, αποδοτικά για να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ο κύριος Λάμπερτ και εγώ συμφωνήσαμε και είπαμε ότι δεν θα ζητήσουμε ε, διαδικασία πρώτης ανάγνωσης. Ε, τα προβλήματα είναι πολύ περίπλοκα, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή πρέπει να προσπαθήσουμε να επεξεργαστούμε ένα χρονοδιάγραμμα όπου αν τηρηθεί ενδέχεται να έχουμε καταλήξει στο τέλος του 2012. Και το λέω αυτό γιατί το χρονοδιάγραμμα δεν θα αποτύχει αν αποτύχει με υπετιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά αν συμβεί του Συμβουλίου. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να συστήσω να ληφθεί μία απόφαση χωρίς να έχει διευκρινιστεί η, ε, ο μέσο πρόθεσμος ε, η μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση. Δεν θα γίνει αυτό που έγινε το 2006, γιατί αν τελικά υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές προτάσεις του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν για το μεσοπρόθεσμο προεπολογισμό την χρηματοδότηση, αυτό ε, θα σημαίνει ότι δεν θα αποφασίσουμε για μικρά και αμεληταία, αλλά θα αποφασίσουμε για μια νέα δομή της ε, πολιτικής συνοχής. Κατόπιν τούτου, εγώ που δεν είναι δεν μπορώ να προτείνω να δεσμευτούμε ήδη τώρα ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012. Όχι. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν. Η Κομισιόν, με την απέραντη σοφία της, βεβαίως πάρα πολλά πράγματα, τα ε, ρύθμισε με απλό τρόπο και μπορεί κανείς να ανακουφιστεί και να πει πάρα πολύ ωραία ε, όλα όσα υπάρχουν, θα, όλα είναι σημαντικά θα υπάρχουν στον κανονισμό και θα ε, εφαρμοστούν με κατεξουδότηση πράξης. Η Κομισιόν θέλει να ε, κρατήσει ακόμα πιο έξω, να απομακρύνει ακόμα περισσότερο το Κοινοβούλιο, το δέχεται κακήν κακός στην νομοθετική διαδικασία η πρόεδρος της ε, Επιτροπής ε, απευθύνθηκε στην νομική υπηρεσία για να ενημερωθεί κατά πόσον όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σωστά ή όχι. Και η πρώτη απάντηση έχει ήδη προκύψει, νομίζω, ή εγώ τουλάχιστον αυτήν την ερμηνεύω ως εξής. Είναι δικαιολογημένο το ερώτημα, μήπως εδώ ε, εκχωρούμε πάρα πολλά. Μήπως θα πρέπει να ελέγξουμε, να δούμε τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτός ο γενικός κανονισμός, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή επιρροή του Κοινοβουλίου ε, σε θέματα επί των οποίων καλούμεθα να αποφάσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η νομική υπηρεσία είπε με απόλυτη σαφήνεια ότι σημαντικές νομοθετικές πράξεις δεν μπορούν να ε, συμπεριληφθούν σε πράξεις κατεξιοδότηση. Ε, άρα δηλαδή τελικό αποτέλεσμα πρέπει να δούμε τι θα περιλαμβάνει αυτός ο γενικός ε, κανονισμός. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο και ε, δεν θα συνεπάγονται μόνο αγώνα και μάχη με την Κομισιόν αλλά και με το Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα τις ε, εταιρικέ συμφωνίες, Όλα αυτά ηχούν πάρα πολύ ωραία και με τις εξηγήσει που έδωσε ο κύριος Μάρτιν σήμερα ηχούν ακόμα πιο ωραία. Όμως για μένα ακόμα, παρόλα αυτά παραμένουν σε πολύ γενικά και αόριστα. Δεν, είναι, δεν έχουν όλα τα κράτη συγκεντρωτική δομή και δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το κατά πόσον θα μπορέσουν να διαπραγματευτούν και οι περιφέρειες. Κατά την άποψή μου αυτό εκρεμεί. Και φτάνω τώρα σε ένα σημαντικό στοιχείο στην ευελιξία και τις ποσοστώσεις. Θεωρώ ότι δεν είναι αιτιολογημένο στον γενικό κανονισμό αλλά και στους κανονισμούς των ταμείων εξακολουθούν να αναφέρονται ποσοστώσεις και ποσοστά και κατ' ουσίαν πρέπει κανείς ε, να ελέγξει κατά πόσο προσθέτοντας τα ποσοστά ε, μήπως ξεπερνάμε και το 100% και φτάνουμε στο 116%. Υπάρχει μόνο ευελιξία και επειδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πάρα πολλές περιφέρειες δεν υπάρχει καθόλου η εγγύηση ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε με την ε, πολιτική της συνοχής και με την ευρωπαϊκή στρατηγική του 2020, κατά πόσον όλα αυτά καλύπτουν τις ανάγκες των περιφερειών. Την ε, προηγούμενη εβδομάδα έκανα την ερώτηση αυτή, την ώρα των ερωτήσεων με την Επιτροπή. Ε, μου είπαν ότι δεν είναι και δικαιολογημένη ερώτηση. Εγώ διαφωνώ, ότι βρίσκω πολύ καλή. Ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε, και σωστό είναι αυτό, ότι σε καμία περιφέρεια δεν υπάρχει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 100%. Όμως, ε, κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να συζητήσουμε για το κατά πόσον η ε, προσέγγιση που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή είναι η σωστή για να επιτύχουμε τους στόχους κλιματικής αλλαγής. Ε. Γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει να ξανακουβεντιάσουμε. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα της απλούστευσης. Ίσως εγώ να είμαι πολύ μεγάλο χρονικό ε, διάστημα στο Κοινοβούλιο. Ξέρω όμω τι σημαίνει έλεγχο των προπολογισμών και αυτά που περιλαμβάνει ο κανονισμός δεν θα συμβάλλουν στην απλούστευση, αλλά φαίνεται ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. <clears throat> Νομίζω λοιπόν το Κοινοβούλιο υποσχέθηκε ότι πρέπει να πλουστεύσουμε. Πρέπει βέβαια να υπάρχει λογικός έλεγχος και καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αυτά πράγματι θα πρέπει ε, να ε, αναφέρουμε στο λάβαρο που θα υψώσουμε. Όσον αφορά την ερεσιμότητα θέλω να πω ότι η δική μου η ε, πολιτική ομάδα απορρίπτει την μάκρο ερεσιμότητα ή επιλεξιμότητα. Έχουμε το παράδειγμα της Ελλάδας και είδαμε τι γίνεται με την Ελλάδα. Συστήθηκε Task Force, ομάδα κρούσης, για να υπάρχει καλύτερη χρήση, αποδοτικότερη των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Και παράλληλα όμως λέμε ότι όταν θα έρθει η επόμενη περίοδος, αυτά τα κονδύλια δεν θα μπορούν να εκταμιευτούν γιατί δεν τηρήθηκαν τα κριτήρια. Και εδώ κάνω το εξή ερώτημα. Ε, τότε η Κομισιόν ε, πότε θα περάσει σε αυτή τη μακροεπιλεξιμότητα ίσως όταν ε, δεν θα τηρούνται τα κριτήρια κατά 0,5-3-5%. εγώ εξ όσων γνωρίζω αυτή τη στιγμή τα κριτήρια του Συμφώνου ε, Σταθερότητας, ε, τα κριτήρια αυτά πληρώνονται μόνο από το Λουξεμβούργο και τη Φιλανδία. Άρα δηλαδή τελειώνει αυτή η πολιτική, πάβει να υπάρχει. Θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Όσον αφορά τώρα το θέμα της ε, αστικής ε, διάστασης, της διάστασης του αστικού ιστού. Εγώ τις προτάσεις της ε, Κομισιόν τις θεωρώ ότι οι προτάσεις αυτές μας επαναφέρουν στα παλαιότερα εργαλεία και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί κάτι διαφορετικό όσον αφορά ε, την ε, αστική βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά είχα να πω. Ο κύριος ε, Λάμπερτ πρέπει και εκείνο να πει κάτι. Την επόμενη φορά ας ξεκινήσει εκείνος και τότε μπορεί να μιλήσει εκείνος περισσότερο. Εγώ αυτά είχα να πω. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε και αρκετή ύλη για συζήτηση για τους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βανίστελ Ρόι, αλλά προηγουμένως ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Αλφόνση δέχτηκε να γίνει συγητής για το να βληθεί η έκθεσή του μάλλον. Άρα μπορούμε να συζητήσουμε τώρα τη συζήτησή μας αύριο μετά την ψηφοφορία. Ο κύριος Βαν Νίστελ Ρόι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε εδώ δύο εισηγητές. Ε, προσπαθήσαμε να συγχρονιστούμε, να μιλήσουμε με ε, έννοια φωνή, να είμαστε με αρμονική, αλλά δυστυχώς δεν τραγουδάω ε, καλά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλούμε για νέα όργανα και εργαλεία και είπαμε ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε με βάση το άρθρο 5 μια διαδικασία με την Επιτροπή Μεταφορών. Και φυσικά θα πρέπει να προχωρήσουμε και στη διαδικασία και να δούμε ποιο θα είναι, ποια θα είναι η διαδικασία που θα εφαρμόσουμε για τη συνοχή και να διατρανώσουμε ευθύ εξ αρχή τη θέση τη Επιτροπή μα στη διαδικασία αυτή. το σημείο 9, 2,5% και το ανώτατο όριο εξαγωγής από το Ταμείο για πολλές χώρες αυτό το ποσοστό δίνει πολύ περίεργα αποτελέσματα. Και φυσικά θέλουμε να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Γιατί αν έχουμε απρόβλεπτα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα, θα πρέπει να το ξέρουμε πριν, να, να καλύψουμε και αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, για το αποθεματικό, ωραία ακούγεται και συγκινητικά, αλλά ίσως επιτείνει τη, τη γραφειοκρατία και περιπλέξει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση. Θα έχουμε πραγματικά διαγωνισμούς ομορφιάς μεταξύ των διαφόρων σχεδίων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την αιρεσιμότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις. Ας δούμε πρώτα, ας τις μελετήσουμε και μετά να εκφέρουμε τη γνώμη μας. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα εξετάσουμε πολύ διεξοδικά. Αλλά πρώτα να λάβουμε τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος. αν αυτό το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, θα πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε, γιατί περιμένουμε το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ας το δούμε πρώτα και ας μην αυτοσχεδιάζουμε. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε και πώς θα εφαρμοστεί συγκεκριμένα ο κανονισμός ε, στις διάφορες χώρες. Και είναι σημαντικό φυσικά να λάβουμε υπόψη και το ρόλο του Συμβουλίου και τη δική του συμβολή. Σας ευχαριστούμε κυρία Μανέσκου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να ευχαριστήσω ε, θερμά και τους ε, δύο εισηγητές για την προσπάθεια που έκαναν. Ευχαριστώ λοιπόν τους δύο συνεισηγητές για το σχέδιο έκθεσης και να πω ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτηματικά και πολλά αδιευκρίνιστα σημεία για το γενικό κανονισμό. Mm. Εγώ θα περιοριστώ σε ορισμένα από τα θέματα που είναι πιο σημαντικά και θα προσπαθήσω να μην μακρηγορήσω για να έχουν την ευκαιρία να λάβουν το λόγο και άλλοι συνάδελφοι. Καταρχήν, ο περιορισμός του προπολογισμού στο 2,5% του ΕΠ. Αυτό πιστεύω ότι είναι αρνητικό και για τις περιφέρειες και για τις... Ε, ε, και για τα κράτη. Και για τα κράτη, ιδιαίτερα όταν ε, υπάρχει αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των περισσότερων και των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών. Θα πρέπει να συζητήσουμε πιο σχολαστικά και διεξοδικά την κατανομή των επιμέρους κονδυλίων του προπολογισμού. Άκουσα τα σχόλια των συνεισηγητών για το διοικητικό και γραφειοκρατικό άχθος. Δεν νομίζω ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, ικανοποιεί το αίτημά μας για απλούστευση. Εξακολουθεί να είναι περίπλοκη και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο οι νέες προτάσεις όντως απλουστεύουν το γραφειοκρατικό άκτος ή αντίθετα το επιτείνουν. Σε ό,τι αφορά ε, τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης ή σύνδεσης, κυρίως ε, συμβάσεις σύνδεσης, εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και στο περιεχόμενο αλλά και στον τύπο, στην ορολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι τοπικές ε, και περιφερειακές αρχές όντως ε, αναμειγνύονται στον καθορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων προκειμένου να καταρτιστούν αυτές οι συμφωνίες σύνδεσης ή εταιρικής σχέσης γιατί αν δεν λάβουμε υπόψη τα αιτήματα των περιφερειών και αν δεν εισακουστεί και η δική τους γνώμη, δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το στόχο της πολιτικής συνοχής. Ένα άλλο θέμα αφορά τον οδηγό, το εγχειρίδιο για τις συμφωνίες αυτές εταιρικής σχέσης και σύνδεσης η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο τάχθηκαν υπέρ αυτού του οδηγού, αυτού του εγχειριδίου για τη σύνδεση. Όπως το είχα προτείνει στη σχετική έκθεση. Αλλά δεν αναφέρεται πουθενά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει και στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να έχουμε ένα τέτοιο εγχειρίδιο, έναν οδηγό. Και επιμένω σε αυτό. Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφορά τον περιορισμό που επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη για τη θέσπιση ε, εθνικών συμπληρωματικών κανόνων. Είναι αλήθεια ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει τη δυνατότητα κάθε κράτος να αυξάνει το διοικητικό άχθος ε, και να επιτείνει το, το τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Νομίζω ότι αυτό αντιβαίνει στο στόχο της απλούστευσης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνουμε πιστοί στα έθιμά μας και να μην επιτρέπουμε στα κράτη να αυξάνουν το διοικητικό άχθος. Ένα άλλο θέμα αφορά τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό κατά πόσο είναι χρήσιμη αυτή η αιρεσιμότητα. Έχουμε και το διδολογικό κώδικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εταιρική σχέση, την σύνδεση. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ένα σαφέστερο οδηγό ε, και ένα διοντολογικό κώδικα για το πώς θα εφαρμοστεί εμπράκτος αυτή η πρόταση. Okay, thank you very much. Ωραία, ευχαριστούμε. Λυπάμαι γιατί ανακοίνωσα διαφορετικά πράγματα, αλλά πρέπει να πω ότι αύριο θα έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε τον κανονισμό Οπότε τώρα ας παραμείνουμε στα γενικά. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στους υπόμενους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές. Τον κύριο Κουτμάνης πρώτα πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πρέπει να συντομεύω γιατί τελειώνει ο χρόνος. Υποστηρίζω αυτά που είπε ο κύριος Βανίστελ Ρόι. η προσπάθεια που έγινε βασιζόταν σε διαφορετικούς κανόνες συνοχής από ό,τι ισχύουν τώρα. Κάτω από 4,9% των χρημάτων του κονδυλίου αυτού έχουν αφιερωθεί στην πραγματική σύγκληση και συνοχή για τον ανταγωνισμό πολύ λιγότερα. Ακόμη και αν τεχνητά πούμε ότι υπάρχει συνοχή και συνδυασμό των προσπαθειών στην Ευρώπη, μόνο αν το πούμε τεχνητά θα μπορέσουμε να το θεωρήσουμε επιτυχία. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι λοιπόν προσπάθησε ένα καινούριο πρόγραμμα να το καλύψει κάτω από τον τίτλο «Συνοχή». Η τωρινή πρόταση της Κομισιόν σήμερα είναι σαφής, δηλαδή να βοηθήσει χώρες με προβλήματα για συγκεντρωτικό έλεγχο και διαχείριση. Αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό στην πράξη. Θα είναι κάτι που ιδιαίτερα δύσκολο για την Κομισιόν. Αν δούμε πώς γίνεται, πώς εφαρμόζεται η περιφερειακή συνεργασία θα δούμε ότι τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Είναι ο χαμηλότερος δυνατός κοινός παρονομαστής που εφαρμόζεται. Πολύ δύσκολο λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα. Δεν αφορά μία χώρα, αλλά πολλές. Και η διασύνδεση όλων αυτών των προβλημάτων μεταξύ όλων των χωρών είναι κάτι το σχεδόν αδύνατο. Θα μπορεί, δηλαδή να καταλήξουμε στην ίδια χαμηλή ποιότητα για όλους. Ε, τότε όμως δεν θα το δεχτούν οι πολίτες γιατί παίρνουμε χρήματα από την κλασική, την παλιά συνοχή και τα βάζουμε σε αυτό το πρόγραμμα που μπορεί να έχει αυτό το αποτέλεσμα. Άμα δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ δύο οδικών συστημάτων, δύο διαφορετικών χωρών, πώς εμείς θα τα συνδυάσουμε με το ζόρι, δεν γίνεται. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει, διότι στις αρχές του χρόνου the things has to be still to The 50... Είδαμε ότι 51% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν από τον μηχανισμό αυτό ήταν αρνητικά, είχαν αρνητικά σε επιπτώσεις και μόνο το 49% ήταν θετικά. Άρα δεν μπορούν να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα με την ίδια ταχύτητα από όλες τις χώρες. Διότι τελικά καταλήγουμε σε 3,5 με 4 φορές μεγαλύτερες διαφορές από ό,τι πριν. Στο επόμενο MFF λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Το 2018 ή 20 θα τα σκεφτούμε αυτά. Τέλος. Όσοι διάβασαν την έκθεση του καθηγητού Μπάρκερ θα θυμούνται ότι προβλεπόταν μία περίοδος υποχρεωτικής πληροφόρησης των από τις χώρες μέλη που δεν αφορούσε μόνο το ρυθμό απορρόφησης αλλά έπρεπε οι χώρες να χορηγήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις, αποτελέσματα των προγραμμάτων δεν τα χορήγησαν αυτά τα στοιχεία όμως. Διάβασα δύο-τρεις μελέτες της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακών και καταλαβαίνω ότι πρέπει τα συμβόλαια μεταξύ μιας χώρας και κομισιών να προβλέπουν την υποχρεωτική αυτή πληροφόρηση. Όχι μόνο ποσοστά, αλλά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Γιατί έχουν χορηγηθεί πολλά κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία σε μερικές χώρες και τώρα πού καταλήγουμε. Αναγκάζεται η Κομισιόν και το Δουνουτού να καταργήσουν τις επιχορηγήσεις αυτές. Ή δίνουν τα λεφτά στους έξυπνους που φεύγουν από τη χώρα, βάζουν τα λεφτά τους σε τρίτες τράπεζες και δεν μπορεί να κάνει τίποτα ούτε το Δουνουτού ούτε η Κομισιόν. Αυτά τα θέματα λοιπόν στη νέα αυτή πολιτική πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά με βάση την πραγματικότητα. Και αν δεν απαντηθούν αυτά εκ των προτέρων δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε τίποτα το θετικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικέ γενικές γραμμέ να σα αναφέρω. Καταρχήν, τι προβλέπει δημοσιονομικά αυτό το πρόγραμμα γενικά. Ξέρω ότι μερικά κράτη-μέλη στο Συμβούλιο το καταπολεμούν. Ξέρουμε ότι είναι όμως Μπορεί να είναι προκλητικές και δύσκολες οι ερωτήσεις αυτές, αλλά είναι απαραίτητο να απαντηθούν. Πρώτον, συνδυασμός των ταμείων. Η συνέργεια των διαφόρων αναπτυξιακών ταμείων είναι κάτι το θετικό αν θέλουμε να καταλήξουμε κάπου. γιατί έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της απλής πολιτικής συνοχής προς ένα πραγματικά εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης να βοηθήσουμε προσωρινά τις περιφέρειες που έχουν δυσκολίες ώστε να μπορέσουν με βάση τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανέλθουν σε καταστάσεις ευημερίας. Υπάρχω, έχω όμως και δύο απορίες. Αυτές οι λεγόμενες ενδιάμεσες περιφέρειες διαρθρώνονται με βάση ορισμένους ρυθμούς συγχρηματοδότησης προοδευτικά μειονόμενους, αλλά το θέμα της ελαστικότητας δεν τις αφορά αυτές τις ενδιάμεσες περιφέρειες. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται και σε αυτές να εφαρμοστεί κάποια ελαστικότητα. Έπειτα, κάτι άλλο που είναι ενδιαφέρον, αυτό το άνοιγμα που λένε στην περιφερειακή ανάπτυξη που να μπορέσει να επιτρέψει πιο αποτελεσματικά προγράμματα. Αυτό καλό αλλά τα νησιά, οι νησιωτικές περιοχές και οι ορεινές περιοχές φαίνεται ότι ξεχάστηκαν γιατί μιλάνε απλώς για περιοχές με λιγότερο πληθυσμό. Τέλος, αν θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά, νομίζω ότι, νομίζουμε ότι πρέπει να στηριχθεί αυτή η πρόταση των πραγματικών αποτελεσμάτων που πρέπει να αναφέρονται. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν ε, θέλησε να σεβαστεί αυτό το αίτημα απλοποίησης και γι' αυτό προτείνει αναλογικότητα των διαδικασιών ανάλογα με τον κίνδυνο που εμπεριέχουν τα προγράμματα. Σωστό μεν είναι αυτό, αλλά θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες για να μην καταλήξουμε τελικά σε λάθη. Περισσότερες λεπτομέρειες. Και τέλος τέλος, το πιο λεπτό σημείο, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα εδώ βλέπουμε πολλές φορές ότι η εφαρμογή των κοντιλίων του Ταμείου Συνοχής ακόμη και σε πολύ δύσκολες δημοσιονομικές καταστάσεις μπορεί να έχει αποτελέσματα όπως είδαμε στην Ελλάδα. Για αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Αυτό θα ήταν μεγάλο λάθος. Τουλάχιστον θα ζητούσαμε η αιρεσιμότητα αυτή να εφαρμόζεται εφόσον έχει αποδειχθεί ότι οι μακροοικονομικά προβλήματα θέτουν σε κίνδυνο την απορρόφηση των προβλημάτων. Αν όπως στην Ελλάδα φανεί ότι υπάρχει τέτοιο πρόβλημα τότε να διατηρηθεί ο υπάρχον μηχανισμός αλλά να, να μην κόβονται αυτόματα τα κονδύλια γιατί έτσι θα χειροτέρευε η κατάσταση αντί να βελτιώνεται. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βλάσακ. Would you please take the floor? Θέλετε παρακαλώ να λάβετε το λόγο αν έχετε την ευγενή καλοσύνη. Κύριε Βλάσακ, τον λόγο, τον λόγο, τον λόγο. Όχι, τότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Κορνιλία Έρνστ. Ε, είμαι σκιώδης συγγήτρια και θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα ε, να αναφέρω τη θέση μας. Ε, κοιτάξτε, όσον αφορά το πολιτές χρηματοδοτικό πλαίσιο, είναι απόλυτα σαφές. Υπάρχουν πολλές αντιφάσκουσες απόψεις για το κατά πόσον το ύψος του του πλαισίου αυτού είναι αποδεκτό και κατά πόσο στηρίζεται από τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ε, κατά τα άλλα, όσον αφορά τα κυλιόμενα ταμεία, αυτό το βρίσκουμε πάρα πολύ καλό. Σήμερα είχαμε και πρόγευμα εργασία και συζητήσαμε για το θέμα αυτό και κατέστη σαφέ ότι σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να εργαστούμε πάρα πολύ καλά. Ε, πρέπει όμω να προσέξουμε να μην υπάρχουν ε, επικαλύψει με το ESF. Τώρα, για τη κατεξουσιοδότηση πράξη. συμφωνώ με την Κωνσταντσα, ε, πράγματι και εδώ πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα διεξοδικά να δούμε αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Γιατί υπάρχουν ε, πολύ σημαντικά θέματα που πρέπει να αποφασιστούν ε, και δεν θεωρώ γιατί όλα αυτά πρέπει η Κομισιό να τα κάνει μόνη της. Γνωρίζω όμως ε, πολύ καλά ότι έρχεται αντίδραση από το Συμβούλιο. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να επανελέγξουμε το θέμα των κατοξιδότηση πράξεων. Για τις ποσοστώσεις λέω τραγικό. Είναι πάρα πολύ αυτό και δεν είναι σαφές ε, κατά πόσο μπορούμε να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία είναι και λογικά. Αν δούμε την ενεργειακή απόδοση, πάρα πολύ ωραία αυτά που λέγονται, όμως έτσι όπως έχουν διατυπωθεί δεν είμαι καν σίγουρη κατά πόσο είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Γιατί ε, υπάρχουν και πράγματα που δεν χρήζουν ενίσχυσης. Υπάρχουν και οι λόγοι γιατί. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο ESF ε, σε σχέση με τον ΕΦΡΑ το 20, δίνει 25% στις λιγότερο αναπτυγμένες ε, και ένα 40% ε, ε, στις ανεπτυγμένες. Πώς εξηγούνται αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Ερεσιμότητα, μακροοικονομική ερεσιμότητα, εμείς την απορρίπτουμε. Και θέλω να επισημάνω το εξής, εξάντε ερεσιμότητα. Αυτό έχει πάρα πολύ καλό. Όμως, έχοντας δει όλα αυτά τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα καταλήγω ε, στο ότι τα εμπόδια είναι πάρα πολύ ψηλά και για χώρες που δεν έχουν ε, τόσο ε, ανεπτυγμένη διοικητική δομή όπως η Γερμανία, το Βέλγιο ή άλλες χώρες, σίγουρα θα έχουν πρόβλημα. Όσον αφορά στο απόθεμα απόδοσης να καταργηθεί, λέω, γιατί έτσι μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο ο προϋπολογισμός. Ε, όσον, όσο προς την, ε, όσον αφορά στην ε, ε, διασύνδεση της Ευρώπης, ελέγχθησαν ορισμένα πράγματα, δεν μου είναι απόλυτα σαφή και στη τελική ανάλυση ε, επιδεινώνεται το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Αυτή είναι μέχρι τώρα η άποψή μας. Σα ευχαριστούμε κύριε Έρνστ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σύντομη αντίδραση. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ θερμά όλους τους ομιλητές για τα σχόλιά τους ε, στον κανονισμό. Βρισκόμαστε στην αφετηρία μια πολύ σημαντική διαδικασία ανταλλαγής απόψεων. Και μια και θα έχουμε και δεύτερη ευκαιρία αύριο για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Προτιμώ να επανέλθω αύριο στις πιο σημαντικές λεπτομέρειες. Τώρα θα σχολιάσω ορισμένα από τα θέματα που επισημάνατε. Η απλούστευση, η απλοποίηση ήταν κάτι που επισήμαναν πολλοί ομιλητέ. Αυτό είναι σημαντικό μέλημα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την εκπόνηση της πρότασης. Γνωρίζουμε πόσο κόπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απλούστευση και είναι σημαντικό αυτό το θέμα και για τους ενδιαφερόμενους αλλά και για τα κράτη-μέλη. Αλλά είναι προς το συμφέρον και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια τέτοια απλούστευση. Θέλουμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα και να μάθουμε κάποια μαθήματα όπως έγινε και στη διαδικασία για τα σχέδια που παράγουν εισόδημα. Και έχουμε και κάποιες καινοτόμες ιδέες, απλουστευμένο κόστος ε, σε κοινά σχέδια δράσης και προσφέρουμε δυνατότητα για μια ναι, ναι, νέα ναι. προσέγγιση στα εφαρμοστικά προγράμματα, αλλά και σε άλλους τομείς. Πάντως, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταθέσουμε ένα πακέτο δράσεων, μια δέσμη δράσεων, για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με την εφαρμογή με τρόπο που να είναι θετική για τους δικαιούχους. Φυσικά θα πρέπει να γίνουν κάποιες δράσεις και στα κράτη-μέλη για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί και εμπράκτος το ρυθμιστικό πλαίσιο, το κανονιστικό πλαίσιο. Γι' αυτό και με κάποιες διατάξεις ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν δράσεις που θα καταλήξουν σε αυτά αποτελέσματα μετρήσιμα. Σε ό,τι αφορά τις και τις εφαρμοστικές πράξεις, όπως διαπιστώσετε, στον κανονισμό υπάρχει πληθώρα μνήων για το δευτερογενές επίπεδο της νομοθεσίας, δηλαδή της κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικές ε, πράξεις. Η συνθήκη της Λισαβόνας αντικαθιστά την ε, επιτροπολογία που είχαμε παλιά. Έχουμε προβεί σε μια αξιολόγηση της νέας κατάστασης και νομίζω ότι έχουμε λιγότερους πια λεπτομεριακούς κανόνες μέσω των ε, κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων. Πολλές διατάξεις του ε, ισχύοντος κανονισμού έχουν ε, περιληφθεί και στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως θα πρέπει να γίνει ε, μια προσεκτική εξέταση, γιατί πρόκειται για ένα νέο στοιχείο και να δούμε πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και ποιος είναι ο σωστότερος τρόπος. Ό,τι αφορά το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, και εκεί θα συνεχιστεί πολύ σημαντική συζήτηση για το κατά πόσο αυτό θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή όχι. Πάντως ε, κατανοούμε τον προβληματισμό σας και θέλουμε να έχουμε την ευκαιρία για πιο διεξοδική συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση και ε, μία των ποσοστώσεων. Σημεία αφετηρίας εδώ είναι ε, η έννοια της συγκέντρωσης και η σημασία αυτής της έννοιας. Αυτό είναι και ο μύθο αριάδνη ε, των προτάσεών μα. Θέλουμε η πολιτική να γίνει πιο αποτελεσματική και εφαρμόζουμε διάφορου τρόπου για να το πετύχουμε αυτό. Η συγκέντρωση των κονδυλίων είναι ένα τρόπο, γιατί από την αξιολόγηση που διεξήγαμε καταλάβαμε ότι ο κατακαιρματισμό των κονδυλίων αποδυνάμωσε την αποτελεσματικότητά του. Και αυτό σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της πολιτικής του 2020 και τις προσπάθειες να είναι πιο αντικειμενικές αυτές οι προτεραιότητες, για να δούμε τι γίνεται πραγματικά με τα κονδύλια, πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια, πώς είναι δυνατόν να, να διοχετεύεται τέτοιο πακτολός χρημάτων και να μην είναι απτά τα αποτελέσματα. Θέλουμε ε, να ε, χρηματοδοτήσουμε σχέδια που πραγματικά έχουν απτά αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι πιο αποτελεσματικά θα είναι τα σχέδια όταν εφαρμόσουν μια συγκέντρωση των κονδυλίων και αναζητούμε ε, μηχανισμούς για να το επιτύχουμε. Ε, για το Περιφερειακό Ταμείο νομίζω ότι δικαιολογείται μια τέτοια προσέγγιση της συγκέντρωσης, αλλά χρειαζόμαστε και πάλι μια πιο λεπτομεριακή προσέγγιση για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Αυτό δεν σημαίνει μηδενική ελαστικότητα, γιατί ακόμη και αν πάρουμε τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές, από το 80% της χρηματοδότησης επικεντρώνεται σε τρεις περιοχές, ακόμη και εκεί υπάρχει δυνατότητα εντός αυτών των τριών περιοχών να αποφασιστεί ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση των κονδυλίων. Το 20% απλώς των ανανεώσιμων είναι ένας στόχος που θα πρέπει να τηρηθεί και υπάρχει το 20% που δεν καλύπτεται, αλλά υπάρχει ελαστικότητα και εξορισμού. Αν θέλουμε συγκέντρωση των κονδυλίων, θα πρέπει να περιορίσουμε την ελαστικότητα. Αυτά προς το παρόν, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι κάλυψα κάποια κεντρικά σημεία, σίγουρα δεν τα εξάντλησα. Αύριο θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία για να συνεχίσουμε τη συζήτηση και αύριο θα σχολιάσω τα υπόλοιπα σημεία. Ευχαριστούμε κύριε Μάρτιν, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίαση και τις παρατηρήσεις σας. Πριν να κηρύξω το συνεδρία σας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα συνεχίσουμε με το Γενικό Κανονισμό, θα ψηφίσουμε και μετά τις ψηφοφορίες θα ακούσουμε τους συνεισηγητές. Κατόπιν θα γίνει συζήτηση και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τους υπόλοιπους κανονισμούς. Αυτά ως προς την δημόσια συνεδρίαση. Παρακαλώ τους συντονιστές να παραμείνουν στην αίθουσα για την συνεδρίαση των συντονιστών.